Καλημέρα σα. Σας καλωσορίζω εγκάρδια στο σημερινό ολοήμερο εργαστήριο μελέτης με θέμα το αστικό δίκαιο και τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων, όσου έχουν έρθει και ελπίζω ότι στο μεταξύ θα έρθουν και άλλοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και καλωσορίζω και τον εκπρόσωπο της ε, Ιρλανδικής Προεδρίας, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, καλωσορίζω τους ευρωβουλευτές, καθώς και όλους τους εμπειρογνώμονές μας που θα λάβουν μέρος στη σημερινή συνεδρίαση και θα μας παρουσιάσουν διάφορες πτυχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Η σημερινή συνεδρίαση περιστρέφεται γύρω από το καθόδε ζήτημα το κατά πόσο οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνουν πραγματικά την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Φυσικά η απάντηση στην ερώτηση αυτή δεν είναι απλή. Γιατί έχουμε το άνοιγμα των συνόρων, την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και χάρη σε αυτό πολλοί Ευρωπαίοι μετακόμισαν, άλλαξαν τον τόπο διαμονής τους, άλλαξαν την οικογενειακή τους κατάσταση, παντρεύτηκαν σε άλλη χώρα, βρήκαν δουλειά σε άλλη χώρα. Οπότε από αυτή την άποψη η απάντηση φαίνεται απλή. Βέβαια, στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης προσώπων ανακύπτουν πολλά νομικά ζητήματα που ταλανίζουν μερικές φορές τους Ευρωπαίους πολίτες και πολύ συχνά δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε σήμερα, ε, οι ευρωπαϊκοί πολίτες ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα και μερικές φορές δεν μπορούν καν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τα νομικά τους δικαιώματα. Πώς θα συμβάλλουμε λοιπόν ε, προκειμένου να τους διευκολύνουμε να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτό θα είναι το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης, του σημερινού εργαστηρίου μελέτης. Θα έχουμε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Για μας είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή για να ανταλλάξουμε απόψεις με ανθρώπους που έχουν αρμοδιότητες παρόμοιες για τα θέματα αυτά. Ελπίζω λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τα κοινοτικά θεσμικά όργανα προκειμένου να μας υποβάλουν τις ε, επόμενες νομοθετικές τους προτάσεις για θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής συνεδρίασης και αυτή είναι η προσδοκία και η ευχή μας. Θα ήθελα ε, να ζητήσω εκ μέρους του κυρίου Λένε, του Προέδρου Τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγγνώμη για την απουσία του, αλλά δυστυχώς ε, η καιρή και το κρύο ε, μερικές φορές ε, βοηθούν την εξάπλωση της γρήπη ή άλλων ασθενειών και πολλοί βρισκόμαστε δυστυχώς ασθενεί. θα ήθελα πάντως να, να ευχηθώ στον κύριο Λένε ταχύ ανάρρωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον καθηγητή Κιον Λένερτ, τον αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκή Ένωση, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του και να του δώσω το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά ως αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που έχω την ευκαιρία να μιλήσω σε αυτή την έγκριτη ομιγύρη και να σας ενημερώσω για τις τελευταίες ε, εξελίξεις της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για θέματα αστικού δικαίου και ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια πολύ συχνά χαρακτηρίστηκε ως η πέμπτη ελευθερία, δηλαδή η ελευθερία που εξασφαλίζει το ελεύθερο δικαίωμα διακίνησης ε, σε οικονομικά ενεργούς πολίτες. Οικονομικά λοιπόν ενεργοί πολίτε ήδη έχουν δικαίωμα ελεύθερη διακίνηση από το 1950. Αυτή είναι η βάση τη εσωτερική αγορά. Και αυτή είναι η ιστορία που έχουμε ακούσει πολλές φορές για την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Οι οικονομικά όμως ανενεργοί ενεργοί πολίτες μπορούν να διακινούνται μόνο εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Οι δύο βασικές προϋποθέσεις της ελεύθερης αυτής διακίνησης είναι να έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και ταυτόχρονα να καλύπτονται από ασφάλεια υγείας. Η πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ επισημαίνει ότι πέραν της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια αποτελεί και μια νομική κατάσταση για τους πολίτες των χωρών μελών και τα εθνικά μέτρα που στερούν de jure ή de facto αυτοδικαίως ή εμπράκτος από τους Ευρωπαίους πολίτες αυτό το καθεστώς, το νομικό καθεστώς ε, της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και τα συμπαρομαρτούντα με αυτό δικαιώματα. Τέτοια εθνικά μέτρα λοιπόν που ακυρώνουν αυτό το δικαίωμα αντιβαίνουν και στο ενωσιακό δίκαιο. Βλέπετε λοιπόν ότι παρόλο που οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή θα γίνει κυρίως ε, περιστρέφεται γύρω από την ελεύθερη διακίνηση μεταξύ των κρατών μελών, δεν περιορίζεται πια σε αυτή την ελεύθερη διακίνηση μόνο εντό των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν καταστάσεις που εκ πρώτης όψεως ε, ακόμη και εσωτερικές ε, καταστάσεις ε, που περιορίζονται σε ένα κράτος μέλος εμπίπτουν ε, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Και θα ήθελα ε, με πολύ συναπτικό τρόπο, μια και μας πιέζει ο χρόνος, να σας δώσω τρία σχετικά παραδείγματα. Η πρώτη περίπτωση είναι η περίπτωση Ρουίς Σαμπράνο. Πρόκειται για την περίπτωση ενός Κολομβιανού ε, υπηκόου και τη σύζυγου του που είναι παράνομη μετανάστες, στο Βέλγιο έχουν έρθει με το παιδί τους που έχει η ηθαγένεια και από τη στιγμή που βρέθηκαν στο Βέλγιο έκαναν και δύο ακόμη παιδιά. Οπότε με βάση το τότε ισχύο δίκαιο ε, του Βελγίου για την ηθαγένεια. Αυτά τα δύο τελευταία παιδιά, τα δύο παιδιά που γεννήθηκαν στο Βέλγιο, απολαμβάνουν την βελγική ηθαγένεια. Θα μπορούσαν να έχουν και Κολομβιανή ηθαγένεια, μια και δεν έκαναν τη σχετική δήλωση όμως ε, στο προξενείο της Κολομβίας. Τα δύο τελευταία παιδιά του ζεύγου είναι Βέλγοι, δηλαδή Ευρωπαίοι πολίτες. Το Βέλγιο αρνείται όμως τον πατέρα των παιδιών, γιατί η μητέρα έχει εξαφανιστεί πια ε, από τη δικογραφία για λόγους άγνωστος προς το ΔΕΚ, γιατί τα πραγματικά περιστατικά είναι γνωστά μόνο στα εθνικά δικαστήρια. Παρ' όλα το Βέλγιο λοιπόν αρνείται να χορηγήσει στον πατέρα άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Το Βέλγιο δηλαδή προτίθεται να απελάσει τον Ρουί Σαμπράνο προς την Κολομβία. Μια και όμως ο, ο Ρουί Σαμπράνο, ο πατέρας των παιδιών, η συνέπεια αυτής της απέλασης θα είναι εκδίωξη και των παιδιών από την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, γιατί πια ο Λούις Αμπράνο δεν θα μπορεί να είναι νόμιμος μεταράστης σε κανένα άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν, ε, η, αυτός ο εκτοπισμός δύο ε, παιδιών που είναι Ευρωπαίοι πολίτες προς μια τρίτη χώρα, την Κολοβία, ουσιαστικά στερεί από τα παιδιά αυτά από τα δικαιώματα που είναι συναφή με, τη, με την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι Βέλγοι που διαμένουν στο Βέλγιο. Αλλά η απόφαση του κράτους ε, της ηθαγένειάς τους, του Βελγίου, να στείλουν τον πατέρα τους που είναι Κολομβιανός επίσης στη χώρα, ουσιαστικά στερεί από τα παιδιά αυτά, de facto, τα δικαιώματα που είναι συναφή με την ε, βελγική τους ηθαγένεια, με την ηθαγένεια μιας χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν είναι μια επιχειρηματολογία που είναι σχετικά περιοριστική, όπως δείχνει η επόμενη ερώτηση ή ε, μια επόμενη υπόθεση του ΔΕΚ, η υπόθεση της κυρίας Μακάρθη. Η Σάρλι Μακάρθη έχει διπλή ηθαγένεια, Ιρλανδική και Βρετανική. Όλη της τη ζωή την έζησε στο Ηνωμένο Βασίλειο και ποτέ δεν αξιοποίησε ή δεν άσκησε το δικαίωμα ελεύθερη διακίνηση μεταξύ των χωρών μελών. Παντρεύεται λοιπόν έναν τζαμαϊκανό υπήκο, που είναι λάθρομετανάστης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει λοιπόν η κυρία Μακάρθη, όπως και ο Λουίς Αμπράνο, θα, θα ήθελα να λάβω άδεια εργασίας για το σύζυγό μου. Ή αν θέλω να συζήσω μαζί του θα πρέπει να φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε το δικαστήριο λέει όχι. Παρόλο που για να έχει κανείς μια αξιοπρεπή οικογενειακή ζωή μπορεί να προτιμάει να μετακομίσει στη Τζαμάικα ε, από, ε, εσείς ως ενήλικα σε, αντίθεση με τα παιδιά στην υπόθεση Σαμπράνο, εσείς μπορείτε να επιλέξετε να ζήσετε είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν η κυρία Μακάρθη μετέβαινε σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει, ο Τζαμαϊκανός σύζυγός της μπορούσε να πάει μαζί της να εργαστεί ή αν πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ε, οδηγίας για τα δικαιώματα του πολίτη για να λάβει την παραμονή πρέπει να είναι οικονομικά ενεργός. Τότε εξασφαλίζεται το δικαίωμα για όλη την οικογένεια να διαμείνει σε άλλο κράτος ε, μέλος. Αλλά απέναντι στο κράτος ε, της ηθαγένης κυρίας Μακάρθη, το Ηνωμένο Βασίλειο, το ενωσιακό δίκαιο δεν, δεν υπερισχύει. Οπότε δεν είναι αναπόδραστη συνέπεια της, του Γραφείου Μετανάστευσης των Βρετανικών Αρχών ότι η κυρία Μακάρθη θα πρέπει να εγκαταλείψει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Γιατί είναι και πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να μεταβεί οπουδήποτε επιθυμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η περίπτωση αυτή δεν καλύπτεται από θέματα της Ευρωπαϊκής Ιθογένειας. Και η κυρία Μακάρθη, σε αντίθεση με τον κύριο Σαμπράνο, της προηγούμενης ε, υπόθεσης δεν ε, δικαιούται παράγω δικαίωμα διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η τελευταία περίπτωση είναι η περίπτωση Ντερέτσι και αφορά έναν Τούρκο υπήκο που διέμενε παράνομα στην Αυστρία, παντρεύτηκε μία Αυστριακή υπήκο και έκανα παιδί που είχε διπλή ηθαγένεια, τυπικότητα, αυστριακή και τουρκική. Ο κύριος Ντερέτσι, στη συνέχεια, ε, υπέβαλε προσφυγή επικαλούμενος στην υπόθεση Σαμπράνο και είπε ότι ναι, το παιδί σου, το παιδί σου εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να αποδειχθεί και αυτό τελικά το αποφασίζει το Εθνικό Δικαστήριο, κατά πόσο η μη χορήγηση δικαιώματος άδειας διαμονής στον κύριο Ντερέτσι θα σημάνει de facto ότι το ανήλικο παιδί του υποχρεούται να εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή επικράτεια. Αυτό λοιπόν που λέω εδώ είναι ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην ομολογία του ΔΕΚ για το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας περιέχουν ένα συστατικό που κρίνει την συμβατότητα των εθνικών μέτρων με το ενωσιακό δίκαιο με βάση τις διατάξεις της Ιθαγένειας, της συνθήκες για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχει ε, κανένα στοιχείο ελεύθερης διακίνησης, όπου οι πολίτες λοιπόν διαμένουν στο κράτος ε, της Ιθαγένειας τους, της εθνικότητάς τους. Παρ' όλα αυτά, μία απόφαση που αφορά ένα μέλος οικογένειας που είναι υπηκός της χώρας μπορεί να έχει τη συνέπεια, ως συνέπεια ε, το την, τον εκτοπισμό, την εκδίωξη ουσιαστικά ενήλικων μελών της οικογένειας ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θερώντας τους de facto από τα δικαιώματα που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε γιατί ίσως έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αντιμετωπίσουν τελείως διαφορετικά το δίκαιο για τη μετανάστευση και την εφαρμογή του δικαίου μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε μέλη της οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι εξελίξεις όμως, όσο σημαντικές και αν είναι, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των συνταγματολόγων και από τη σκοπιά των συνταγματολόγων, δεν θα πρέπει να μας αποσπούν την προσοχή από το γεγονός ότι το βασικό στοιχείο ε, του νόμου για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια είναι η ελεύθερη διακίνηση και το δίκαιο σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση. Αν εξετάσουμε όλες τις υποθέσεις και όλη την ομολογία του ΔΕΚ για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια διαπιστώνουμε ότι 90% των υποθέσεων αφορούσαν την περίπτωση υπηκών μιας χώρας που έχουν μετακομίσει, έχουν μεταβεί σε άλλη χώρα, εργάζονται εκεί, διαμένουν εκεί, εγκαθίστανται ως ανεξάρτητοι εργαζόμενοι και ούτω καθεξής. Και φτάνοντας τώρα στο θέμα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που είναι και το κυρίως θέμα του σεμιναρίου αυτού, φτάνω σε περιπτώσεις, σε υποθέσεις που αφορούν ονόματα οικογενειακά. Γνωρίζετε την περίπτωση του Καρθία Βάλιο. Μία υπόθεση όπου ένας Ισπανός πατέρας και μία Βελγίδα μητέρα έχουν δύο παιδιά από κοινού και τα παιδιά αυτά λαμβάνουν το όνομα του πατοργωνιών με βάση το Ισπανικό δίκαιο. Παίρνουν και το Γκαρθία, το επίθετο Γκαρθία και το επίθετο Βέμπερ και το επίθετο του πατρός και το επίθετο της μητρός. Κατ' εφαρμογή του Ισπανικού δικαίου σε ό,τι αφορά την ονοματοδοσία. Η οικογένεια αυτή όμως διαμένει στο Βέλγιο και το Βέλγιο λέει όχι. Μια και τα παιδιά είναι και Βέλγιοι υπήκοοι, εκτός του ότι είναι και Ισπανοί, θα πρέπει να έχουν μόνο το επίθετο του πατρό. Γιατί αυτό προβλέπει το βελγικό δίκαιο. Και με βάση την ε, παλιά συνθήκη της Χάγης του 31, ένα κράτος μπορεί να θεωρήσει ότι οι πολίτες με τη, με τη διπλή θαγένεια, με πολλαπλή θαγένεια μπορούν να θεωρούνται πολίτες ε, του συγκεκριμένου ε, κράτους εφόσον διαμένουν σε αυτό. Οπότε για, τα, για τις βελγικές αρχές τα παιδιά αυτά είναι μόνο Βέλγοι και εφαρμόζεται σε αυτά το βελγικό δίκαιο για την προσωπική τους κατάσταση δηλαδή. Οι γονείς προσέφηκαν σε βελγικό δικαστήριο. Το βελγικό δικαστήριο παρέπεψε το θέμα στο ΔΕΚ. Το ΔΕΚ αποφάσισε, ε, εκδίκασε το θέμα δίνοντα απόφαση κατά του Βελγίου, λέγοντας ότι μια και είναι ευρωπαϊκό αυτό το θέμα, δημιουργείται ένα σημαντικό πρόσκομα με την επιχειρηματολογία σας λέει το ΔΕΚ στις βελγικές αρχές. Γιατί αν το Βέλγιο θεωρεί ότι τα παιδιά έχουν μόνο την βελγική ηθαγένεια και άρα δικαιούνται να έχουν μόνο το επίθετο του πατρός, τότε η Ισπανία μπορεί να θεωρήσει ότι τα παιδιά είναι μόνο Ισπανοί υπήκοοι. Και άρα έχουν το, το, διπλό επίθετο, το πατρός και της μητρός, που σημαίνει ότι στα επίσημα έγγραφα, τα ισπανικά και τα βελγικά, τα παιδιά αυτά θα είχαν διαφορετικά επίθετα, διαφορετικά ονοματεπώνυμα. Τι θα συμβεί όμω αυτό με την ταυτότητά του, με τα διαβατήριά του, τι θα λένε τα διαβατήριά τους όταν θα ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι από τη στιγμή που κατ' εξαίρεση και το βελικό δίκαιο η επιλογή ενώ, και ενό άλλου επιθέτου πέραν της αυτόματης ε, υιοθέτηση του επιθέτου του πατρό, το Βέλγιο θα πρέπει να επιδείξει ε, μία μεγάλο και να εφαρμόσει αυτή την ε, ελευθερία επιλογής σε περίπτωση που τα παιδιά δεν είναι μόνο Βέλγοι υπήκοοι, αλλά έχουν διπλή ηθαγένεια, έχουν και την Ισπανική ηθαγένεια. Οπότε τα παιδιά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυκλοφορούν με το διπλό επίθετο. Γκαρθία Βέμπερ. Αλλιώς ε, θα δημιουργούνταν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνησή τους. Πάντως ε, με βάση το διεθνό, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει η περίπτωση, περιβόητη περίπτωση περίπτωση Kim Paul. Και μάλιστα εγώ ως ειδικό για το ιδιωτικό διεθνέ δίκαιο θεωρώ αυτή την υπόθεση ακόμη πιο σημαντική γιατί έχουμε μια ολόκληρη γερμανική οικογένεια, γερμανό πατέρα, γερμανή μητέρα, γερμανίδα μητέρα που εργάζονται στη Δανία. Ε, κάνουν ένα παιδί, ένα γιο και η Δανία Ε, σε αντίθεση με τη Γερμανία ή το Βέλγιο, συνδέει την προσωπική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση του προσώπου, όχι με την ηθαγένειά του, αλλά με την συνήθη διαμονή του. Οπότε ισχύει το δίκαιο της συνήθους διαμονής του Γερμανού παιδιού από δύο Γερμανούς πατέρες. Ε, είναι το δίκαιο αυτό το δανεικό δίκαιο. Και το, δανεικό, το δανέζικο δίκαιο ε, αφήνει την ελεύθερη επιλογή του επιθέτου στους γονείς. Οι γονείς αποφάσισαν να λέγεται Γκρίμκιν, Παύλα και μετά το επίθετο της Μητρός. Γκρίμκιν, Παύλα, Πολ. Διπλό επίθετο, πατρός και μητρός. Με βάση την ελεύθερη επιλογή που χορηγεί το δανεικό δίκαιο. Μετά από μια δεκαετία δυστυχώς χωρίζει το ζευγάρι και ένας από τους γονείς επιστρέφει στη Γερμανία με το παιδί και θέλει να γραφτεί στο Μητρό Πληθυσμού, στο Ληξιαρχείο, στο Βέλγιο, στο, στη Γερμανία, συγγνώμη. Και εκεί ο Ληξίαρχος ε, τους λέει το παιδί είναι Γερμανός πολίτης. Ως εκ τούτου το όνομά του θα πρέπει να συμμορφώνεται με την γερμανική νομοθεσία που συνδέει το επίθετο με την, ε, με την ηθαγένεια. Άρα το παιδί θα πρέπει να λέγεται μόνο Γκρίμκιν, όπως ο πατέρας του. Οι δύο γονείς, παρόλο που στο μεταξύ έχουν ε, χωρίσει, έχουν πάρει διαζύγιο, συμφωνούν ότι το παιδί τους θα πρέπει να φέρει το διπλό επίθετο, όπως και στο παρελθόν, και προσφεύγουν στο δικαστήριο. Το Γερμανικό Δικαστήριο θέτει προδικαστικό ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πολύ εύστοχα κατά τη γνώμη μου, ε, επισημαίνει ότι από τη στιγμή που κάποιος νόμιμα αποκτά σε ένα κράτος μέλος μία προσωπική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση με βάση το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο και το ουσιαστικό δίκαιο που καλύπτει, ε, που ισχύει από το από το αρμόδιο κράτος. Τη στιγμή που λαμβάνει αυτό το καθεστώς λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα κράτη, ακόμη και το κράτος μέλος της Ιθαγένειας θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτή την προσωπική κατάσταση που έχει αποκτηθεί νομίμως. Με μόνο μία εξαίρεση που είναι γνωστή στο ιδιωτικό διεθνέ δίκαιο με την εξαίρεση της δημόσιας τάξης. Αλλά η Γερμανία αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε καμία προσβολή της δημόσιας τάξη η διατάραξη της δημόσιας τάξης. Ήταν ένα θέμα μόνο ε, νομικών κανόνων και επιλογής του δικαίου. Το ΔΕΚ είπε ότι δεν είναι θέμα επιλογής δικαίου, είναι θέμα αναγνώρισης μιας προσωπικής ε, νομικής κατάστασης που έχει εκτιθεί νομίμως στο συγκεκριμένο χρόνο, τη στιγμή της γέννησης δηλαδή, όταν το παιδί έλαβε αυτό το διπλό επίθετο. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν τη σημασία που έχει το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο για τους Ευρωπαίους πολίτες και για την ε, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Οπότε είναι πραγματικά αξιέπαινο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οργανώνει σήμερα αυτό το σημαντικό εργαστήριο μελέτης και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που συμμετέχω σε αυτή την εισαγωγική ενότητα. Γιατί ο Ευρωπαίος νομοθέτης με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που είναι και καταλληλότερη για τέτοιου είδους θέματα γιατί πρόκειται για θέματα που αγγίζουν άμεσα τους πολίτες ε, ε καλείται να εγκρίνει αυτούς τους ε, νέους κανόνες και σε επίπεδο εφαρμοστέου δικαίου, δηλαδή διατάξεις τύπου Ρώμης. Και γιατί λέω Ρώμης, γιατί οι πρωτοφυγές προσπάθειες της νομικής ε, Ένωσης για το εφαρμοστέο δίκαιο είναι η συνθήκη της Ρώμης του 1980 που ε, ισχύει στις ενοχές, στις συμβατικές ενοχές. Είχαμε τον κανονισμό Ρώμη 1 και μετά τον κανονισμό Ρώμη 2 για τις έξω συμβατικές ή μη συμβατικές ενοχές. Και έχουμε και μία σειρά κανονισμών για το εφαρμοστέο δίκαιο. Έχουμε τις διατάξεις που ισχύουν για ε, διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό και είχαμε πρόσφατα τον κανονισμό 650 του 2012 που μιλάει για το εφαρμοστέο δίκαιο που ισχύει για, τις, ε, για την κληρονομική διαδοχή και τις διαθήκες ε, τις οποίες θα, μας, θα έχουμε μια παρουσίαση το απόγευμα. Έχουμε όμως και τους αυτοί οι κανονισμοί των Βρυξελών καθορίζουν τη διεθνή δικαιοδοσία των διαδικαστηρίων και την αναγνώριση, τον εκτελεστήριο τίτλο, εξεκουάτορ, θα πρέπει να αναφερθούν αυτοί οι κανονισμοί των Βρυξελών. Και θα ήθελα να χαιρετήσω ιδιαιτέρως και να ποτίσω φόρο τιμής στο αξιόλογο και πολύ ποιοτικό έργο που γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων από ευκαιρία της αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξέλλες 1 που υιοθετήθηκε με μορφή αναδιατύπωση το Δεκέμβριο του 2012 και πολύ πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σε αυτή την αναδιατύπωση λοιπόν του κανονισμού των Βρυξελών βρίσκουμε πολλές νομοθετικές απαντήσεις που σχετίζονται με την ομολογία του ΔΕΚ και που εκδόθηκαν στα πλαίσια του προηγούμενου κανονισμού των Βρυξελών 1. Ο προηγούμενος κανονισμός πριν την αναδιατύπωση ήταν ουσιαστικά τέκνο από κύμα της αρχικής ε, σύμβασης η συνθήκη των Βρυξελών που έχει αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον αρχικό κανονισμό Βρυξέλλες 1. Οι διαπραγματεύσει είχαν γίνει στη δεκαετία του 60 όταν η χώρες του Common Law και η παράδοση του Common Law δεν αποτελούσε τμήμα του του δικαίου του Ιους Κομούνε των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τότε. Είχαμε βέβαια τις ενταξιακές ε, συμφωνίες, αλλά δεν ε, δημιουργούσε πλήρη ένταξη του common law. Και μια πραγματική νομοθετική αναδιατύπωση έγινε μόνο τελευταία αιτία και μάλιστα με πρωτοβουλία ε, και παρότριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Και πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της νομοθετικής διαδικασίας. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο τροποποίησεις του νέου αυτοκανονισμού που σίγουρα θα ε, οδηγήσουν σε περαιτέρω εξελίξεις ε, της νομολογίας του ΔΕΚ. Όχι γιατί η προηγούμενη νομολογία ήταν ε, ανακριβής ή εσφαλμένη, ήταν σωστή με βάση το τότε ισχύον δίκαιο. Το δίκαιο όμως έχει τροποποιηθεί και άρα και η νομολογία θα εξελιχθεί αντίστοιχα. Θα ήθελα να σας παραπέμψω καταρχήν στο άρθρο 1.2, όπου ο νέος κανονισμός προβλέπει εξαίρεση από το Γενικό Κανόνα της Κρεμοδικίας, Λις Πέντενς, με βάση την, τον οποίο ε, το δεύτερο ή τρίτο δικαστήριο που έχει επιληφθεί θα πρέπει να παραπέμψει στο δικαστήριο της πρώτης προσφυγής, που έχει επιληφθεί πρώτο. Γιατί η αμοιβαία εμπιστοσύνη προβλέπει το πρώτο δικαστήριο που έχει επιληφθεί θα κάνει τη σωστή εκτίμηση των κανόνων της διεθνούς δικαιοδοσίας και τα υπόλοιπα δικαστήρια θα το λάβουν αυτό υπόψη. Υπάρχει όμως μια εξαίρεση αυτόν τον κανόνα του Λις Πέντενς της εκκρεμωδικίας και η εξαίρεση αφορά μια συμφωνία σε σύμβαση που χορηγεί αποκλειστική αρμοδιότητα σε ένα δικαστήριο ακόμη και αν έχουμε ένα πρώτο επιλεφθέν δικαστήριο που δεν είναι το δικαστήριο που έχει καθοριστεί στην συμφωνία που χορηγεί αποκλειστική αρμοδιότητα, το δεύτερο δικαστήριο είναι το δικαστήριο που αναφέρεται στη συμφωνία αποκλειστικής αρμοδιότητας. Οπότε το δεύτερο δικαστήριο θα ε, κρίνει την εγκυρότητα της ρήτρας διεθνούς δικαιοδοσίας του, της σύμβασης. Και το πρώτο απελευθεία δικαστήριο θα πρέπει να περιμένει. Αυτή είναι σημαντική εξαίρεση και μια πολύ σημαντική τροπή καμπή στη νομολογία του ΔΕΚ. Και το λέω αυτό σε όσους ειδικού γνωρίζουν την ε, υπόθεση Γκάστερ. Σημαντική τροπή λοιπόν. Το ίδιο ισχύει για τα άρθρα 34, 33 και 34 που με βάση την αλλαγή της νομοθεσίας Γούσου προβλέπει δυνατότητα σε περίπτωση που εκκρεμωδική μία υπόθεση σε ένα δικαστήριο τρίτης χώρας το δικαστήριο του κράτους μέλους που έχει διεθνή δικαιοδοσία με βάση τον κανονισμό Βρυξέλλες 1 παρόλα αυτά παρόλα αυτά θα περιμένει θα αναστείλει τη διαδικασία ε, εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου της ε, τρίτης χώρας. Ιδιαίτερος, αν η απόφαση του δικαστηρίου της τρίτης χώρας αφορά την εκτελεστότητα στο κράτος μέλος στο οποίο έχει ασκηθεί και στο οποίο έχει ασκηθεί προσφύγη. Όλα αυτά δείχνουν ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ο Ευρωπαίος νομοθέτης που μας φιλοξενεί σήμερα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκούν και εκπληρώνουν ε, συμπληρωματικούς ρόλους σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης. Γιατί η αστική δικαιοσύνη είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα, αλλά και η εκ των άνευ προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια που δημιουργεί μια κατάσταση στα κράτη-μέλη η οποία συνδέεται με συγκεκριμένο πλέγμα δικαιωμάτων τα οποία είναι αναφέρετα από το κράτος μέλος. Υποθέσεις ε, Λουίς Σαμπράνο και Μακάρθη. Τα ίδια αυτά δικαιώματα ε, προβλέπουν ελεύθερη διακίνηση και άρα επαφές και τριβές και με άλλα νομικά συστήματα. Οπότε είναι σημαντικό με απόλυτη ακρίβεια και απόλυτη προβλεψιμότητα να γνωρίζουμε ποιο φόρουμ, ποιο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και κατά πόσο οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με τέτοιο τρόπο, νομότυπα, που θα, αν θα αναγνωρίζονται, πώς θα εκτελούνται και υπό προϋποθέσεις και όρους. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα της σημερινής ε, συζήτησης. Το 10 ε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την πρόοδο και τις εξελίξεις των νομοθετικών κανόνων και χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δόθηκε ευκαιρία να σας παρουσιάσω και εγώ μερικές σκέψεις συμβάλλοντας ε, στο εργαστήριο αυτό μελέτης που δυστυχώς δεν θα παρακολουθήσω μέχρι τέλους γιατί σε μισή ώρα έχω άλλη η υποχρέωση κάπου αλλού στις Βρυξέλλες και το απόγευμα πρέπει να μεταβώ στο Λουξεμβούργο, στο δικαστήριο. Πάντως σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά, κύριε Λέναρτς. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ομιλία σας για θέματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και για θέματα που ε, αποτελούν τα αντικείμενα προσφυγής ε, και στο ΔΕΚ. Είναι σημεία που δημιουργούν κάποια προσκόμματα στην ε, απρόσκοπτη, κανονικά θα, όπως θα έπρεπε, λειτουργία και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Και για την επίλυση των προβλημάτων αυτών χρειαζόμαστε ένα, τουλάχιστον μια καλή βούληση. Καλή επίστη και καλή βούληση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λέναρτς. Εγώ είχα την χαρά να είμαι ο εισηγητής στην αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Ε, ήταν τεράστιο αυτό το έργο και μάλιστα και χρονοβόρα διαδικασία. Κράτησε μία διετία, αλλά θα ήθελα να τονίσω την αγαστή συνεργασία που είχαμε με τις Προεδρίες του Συμβουλίου, αλλά και την προθυμία της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να διεκπαιρεώσουμε αισίως τις διαδικασίες για την τροποποίηση του κανονισμού αυτού και το θέμα της αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και την εκτέλεσή τους στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε και πάλι κύριε καθηγητά και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Άλαν Σάτερ που είναι Υπουργός Δικαιοσύνης ε, της Ιρλανδίας και στα πλαίσια της Προεδρίας θα μας αγραφήσει τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας για το αστικό δίκαιο για το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήδη ευθύ εξ αρχή θα ήθελα να σας πω ότι με μεγάλη χαρά έρχομαι εδώ ενώπιόν σας. Θα ήθελα να αναγνωρίσω τη θαυμάσια δουλειά τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης και να αποτίσω φόρο τιμής το πνεύμα συνεργασίας που διαπνέει τις ε, εργασίες της Επιτροπής σας σε αυτόν τον τομέα. Με ειδική χαρά άκουσα την ομιλία του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι η Ιρλανδία ανέλαβε την Προεδρία και εγώ έχω το χαρτοφυλάκιο δικαιοσύνης. Ως δικηγόρος, μία από τις ειδικότητε μου, πέρα από την πολιτική μου ζωή, φυσικά καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου, μια και είμαι υπουργό, αλλά ένας από τους τομείς που με ενδιέφεραν πάντα ήταν ε, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Και όλοι σας αυτοί, ε, όλα τα θέματα τα οποία θα συζητήσετε σήμερα, είναι αυτά που με απασχόλησαν επί 30 χρόνια. Είναι το τομεί όπου και εσωτερικά στην Ιρλανδία θα κάνουμε κάποιες ε, εθνικές μεταρρυθμίσεις ε, σχετικές με τα θέματα που θα συζητήσετε σήμερα. Φυσικά στον τομέα του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου έχουμε κοινό συμφέρον να εξασφαλίσουμε ότι προωθούμε τα θέματα με ομοιόμορφο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προ το συμφέρον των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω με ανυπομονησία, παρά δεν θα μπορέσω να παραστώ σε όλη την συνάντησή σα, γιατί έχω και άλλε υποχρεώσει. να λάβω ένα αντίγραφο της μελέτης για μια συγκριτική ανάλυση ε, για το δίκαιο που διέπει τα θέματα της παρένθετης μητέρας. Εμεί στην Ιρλανδία προσπαθούμε να δούμε τα θέματα της κυδαιμονίας, ε, του ποιο είναι ο γονιός και όλα τα θέματα τα οποία προκύπτουν από την ε, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και ε, τα θέματα που σχετίζονται με τις παρένθετες μητέρες. Επομένως αυτά ειδικά τα κείμενα περιμένω να τα δω μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα για κάποιες από τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ξέρω ότι υπάρχουν προτεραιότητες που μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα και χρειαζόμαστε γι' αυτό όμως την συνεργασία και τη βοήθεια της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Υπάρχουν μία πλειάδα θεμάτων που απασχολούν την Ιρλανδία και την κυβέρνησή μου και στο πλαίσιο της ε, Προεδρίας ε, και εμένα όμως ε, προσωπικά. Κατά τη διάρκεια του πρωινού ε, εξήγησα σε έναν συναδελφό μου ότι κληρονομήσαμε τέσσερα θέματα. Εκείνος μου έλεγε μάλλον ότι κληρονόμησε τέσσερα θέματα, αλλά εγώ 51. Η Ιρλανδική Προεδρία, λοιπόν, θα δώσει ειδική προτεραιότητα στα νομοθετικά μέτρα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Αλλά δεν θα δώσουμε μόνο προτεραιότητα σε αυτά. Εγώ θέλω να εστιάσω στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης και φυσικά εδώ υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα ε, και στον τομέα της, ε, των εσωτερικών υποθέσεων και της μετανάστευσης που μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη και στην α, ε, α, ε, ανάκαμψη. Παραδείγματο χάρη κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων και προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με σκοπό να μην υπάρχουν πλέον οικονομικά κίνητρα για έγκλημα και έμεσα να υποστηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε την νόμιμη οικονομική δραστηριότητα. Ε, με την πολιτική μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία ε, ανάμεσα στην ασφάλεια των συνόρων μας και στην διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστασης, να συμπληρώσουμε το εργατικό δυναμικό της Ένωσης με ανθρώπους με ειδικά προσόντα και πραγματογνωμοσύνη. Αυτό σημαίνει προτάσεις για εδωτερικέ μεταθέσεις και εποχικούς εργαζόμενους. Αυτά θα είναι επίσης στο κέντρο της, των εργασιών της Προεδρίας μας. Στις πολιτικές μετανάστευσης επίσης θέλουμε να τις προωθήσουμε με έναν τρόπο ανθρώπινο, αναγνωρίζοντας τα ατομικά δικαιώματα των ενηλίκων και των ε, πολιτών της Ένωσης. Και άκουσα την, ε, στην ομιλία του Αντιπροέδρου, άκουσα να λέει την πολύ σημαντική ε, απόφαση, την απόφαση Ζεμπράνο. Όταν ανέλαβε υπουργό ε, Δικαιοσύνη, αμέσω μετά ελήφθη αυτή η απόφαση. Και θα εφαρμόσουμε και στην Ιρλανδία την πολύ λογική απόφαση του δικαστηρίου ε, για την υπόθεση Ζεμπράνο. Έχουμε χίλιες σχετικές αιτήσει από άτομα τα οποία προσπαθούν ε, να παγιώσουν το δικαίωμά τους για την κατοικία. Οι αρχέ τη υπόθεση ε, Ζεμπράνου είχαν λοιπόν ε, σημασία και επιπτώσεις και για την Ιρλανδία. Κοιτώντα λοιπόν τώρα την ευρωπαϊκή οικονομία, ε, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πληθυσμό πάνω από 500 εκατομμύρια. Ε, υπάρχουν ενδείξει ανάκαμψη ό,τι αφορά το ρυθμό ανάπτυξη και τι εξαγωγέ εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγαθά και υπηρεσίε. Ε, αυτό στην εσωτερική αγορά και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ένα μερίδιο 20%. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημερινό εμπορικό περιβάλλον είναι και μια ευκαιρία αλλά και μια πρόκληση. Και εμείς ως Προεδρία ε, στην αστική δικαιοσύνη θα εστιάσουμε κυρίως σε αυτά τα μέσα και εργαλεία που μπορούν να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξη και στην ασφάλεια της απασχόλησης. Μία από τις ε, μεγάλες προτεραιότητες μας είναι η πρόταση για να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησης ε, λογαριασμών. Έχουμε 10 ημέρες συνετριάσεων στο Συμβούλιο για να υιοθετηθεί πολύ γρήγορα αυτό το κείμενο. Μία σημαντική πτυχή του είναι ότι αναγνωρίζει μια μεγάλη δυσκολία για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ε, σε οποιοδήποτε διασυνοριακό περιβάλλον. Και με αυτή την πρόταση βρίσκουμε λύσεις όταν κάτι πάει στραβά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Όταν παρέχει κάποιος υπηρεσίες και αγαθά σε ένα άλλο κρατός μέλος και όταν ε, εκείνοι που έχουν παραλάβει αυτά τα αγαθά της υπηρεσίας δεν σε πληρώνουν. Η προτινόμενη αυτή πρόταση έχει σαν σκοπό να μειώσει τον κίνδυνο για τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε διασυνοριακό εμπόριο, διευκολύνοντας την ανάκτηση διασυνοριακών χρεών. Όπως θα γνωρίζετε σίγουρα, ο προτινόμος κανονισμός προβλέπει την ε, δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής διαδικασίας που θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα πιστωτή να εμποδίσει τη μεταφορά ή την απόσυρση των πλουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η στοχη τη πρόταση είναι να διευκολύνει την ανάκτηση διασυνοριακών απαιτήσεων για του πολίτε και τι επιχειρήσει, ειδικά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τη εκτέλεση των ε, ε, δικαστικών αποφάσεων σε εμπορικά θέματα και θέματα αστικού δικαίου όταν έχουμε διασυνορικές ε, διαφορέ. Ένα τέτοιο πιο ασφαλέ περιβάλλον θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των εμπορευομένων, θα ενθαρρύνει περισσότερη διασυνοριακή δραστηριότητα. Σήμερα έχουμε οικονομικ... όλοι αντιμετωπίζουμε οικονομικέ δυσκολίε, σε όλα τα κράτη-μέλη και ακριβώ γι' αυτό η πρόταση είναι πολύ σημαντική. Η πρόταση επίσης ε, καλύπτει ένα κενό που υπάρχει στα σημερινά εργαλεία στον τομέα τη αστική δικαιοσύνη. Γιατί αυτά τα εργαλεία όπως ε, το, η πρόσφατη αναθεώρηση του Βρυξέλλες 1 ε, προβλέπουν την ε, εκτέλεση αποφάσεων αλλά η διαδικασία εκτέλεσης σε αυτή τη φάση διέπεται από διαφορετικά καθεστώτα σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Το πάγωμα των λογαριασμών επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτόν τον τομέα. Για την ουσία του κανονισμού έχουμε σαν σκοπό να εστιάσουμε ειδικά στην επαρκή προστασία του οφηλέτη και να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο περίπλοκη ή τόσο επαχθής, ούτως ώστε να αποτρέπει τους πιστωτές να τη χρησιμοποιούν και να ανακτούν ε, τα, τις οφειλές. Ελπίζω να συνεργαστούμε με την Επιτροπή σας για αυτόν τον κανονισμό. Φυσικά η επιχειρηματική δραστηριότητα ε, ενέχει κινδύνους στην ενιαία αγορά. Όταν έχουμε ε, διαδικασίες αφαιρεγγιότητας διασυνοριακές, θα πρέπει να έχουμε τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες προφανώς. Αυτές οι διαδικασίες όταν χρειάζεται θα πρέπει να μπορούν να βοηθήσουν ε, στη διάσωση ε, βιώσιμων επιχειρήσεων, τίμιων επιχειρηματιών και στην ελάφρυνση ε, πολύ παχθών φόρων που έχουν άτομα λόγω Ενό εμπορικού ε, χρέους, ε, προσωπικού χρέους ή υποθήκης. Η πρόταση τη 12 η Δεκεμβρίου του 2012 από την Κομισιόν για ένα κανονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που να τροποποιεί τον κανονισμό του 2000 για την ε, αφαιρεγκαιότητα ήταν πολύ επίκαιρο. Τον καλωσορίζω γιατί εκείνη τη βδομάδα που ολοκληρώσαμε την προσπάθειά μας στην Ιρλανδία για μια μεγάλη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας μας για την αφαιρεγγιότητα που σκοπό έχει να δώσει στα άτομα μια εναλλακτική λύση στην πτώχευση όταν βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες και να προβλέψει επίλυση, εξοδικαστική επίλυση διαφορών σε περίπτωση που υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στον πιστωτή και στον οφηλέτη με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, ο οποίος είναι ειδικό για θέματα αφαιρεγγιότητας. Το όφελος του κανονισμού που προτείνεται είναι ότι θα επιτρέψει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να, αναγνωρίζεται, να αναγνωρίζονται οι αποφάσεις για την πτώχευση, αλλά θα αναγνωρίσουμε το θέμα επίσης του βασικού κέντρου οικονομικών συμφερόντων ενός ατόμου, αλλά προβλέπει επίσης την αμοιβαία αναγνώριση νέων τρόπων επίλυσης των διαφορών εκτός δικαστηρίου, χωρίς αντιπαράθεση. Προβλέπουμε δηλαδή μία πλειάδα από περιπτώσεις και μπορούμε να αναγνωρίσουμε διάφορες ε, διαφορές ε, και να τις επιλύσουμε με διαφορετικό τρόπο. Ο κανονισμός αυτός λειτουργεί αποτελεσματικά. Ε, Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για εξυγχρονισμό και διευκρίνηση ορισμένων πτυχών του. Ένα παράδειγμα αφορά αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το πού βρίσκονται τα βασικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα του οφειλέτη. και τι μηχανισμούς θα έχουμε ε, για την ε, αφαιρεγγιότητα που δεν είναι επιτόχευση. Ο εξυγχρονισμός αυτών των διαδικασιών θα μας βοηθήσει ούτως ώστε να βάλουμε την οικονομική ανάπτυξη στο κέντρο της ατζέντα μας για την ε, αστική δικαιοσύνη και να ενισχύσουμε την νέα αγορά. Η πρόταση αναγνωρίζει την ανάγκη να ανταποκριθούμε στα σημαντικά προβλήματα υπερχρέωσης που έχουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας, στις πολύ ζωφερές οικονομικές συνθήκες σε ό,τι αφορά τι διαδικασίε αφαιρεγγιότητας που είναι διασυνοριακές, θέλουμε όπου μπορούμε να απομακρυνθούμε από μια προσέγγιση που να αφορά την εκαθάριση κατά την αφαιρεγγιότητα και να εστιάσουμε στη διάσωση και αναδιάρθρωση της επιχείρησης, ε, αντισταθμίζοντας ε, τα συμφέροντα, τα νόμιμα συμφέροντα και τις προτοκίες των πιστωτών και όταν γίνεται δυνατό να μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε οικονομικά κάποιες ε, επιχειρήσεις. Να μην χρειαστεί δηλαδή, να καθαρίσουμε μια επιχείρηση όταν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Οι εξελίξεις ε, και η αλλαγή της διαδικασίας ε, θα απαιτήσει μια ανοιχτή προσέγγιση από τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν ε, κατά τη διάρκεια της ε, διαπραγμάτευσης και ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη όπως και η Ιρλανδία έχουν εξυγχρονίσει τους, την εθνική του νομοθεσία για την αφαιρεγκαιότητα και άλλα κράτη-μέλη είναι στη διαδικασία της, του εξυγχρονισμού στο άτυπο Τζάι του Δουβλίου την περασμένη εβδομάδα, οι υπουργοί είχαν μια ενδιαφέρουσα αρχική συζήτηση για την πρόταση τη Κομισιόν περί αφαιρεγκαιότητα και μπορώ να σα πω ότι υπήρξε θετική υποδοχή από του υπουργού τη πρόταση τη Κομισιόν. Η πρόταση, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Αφαιρεγκαιότητα, είναι προτεραιότητα τη ε, Προεδρία μα και έχουμε προβλέψει έξι ημέρε ε, συνεδριάσεων τη ομάδα εργασία. Ελπίζω να μπορέσουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Η ενίσχυση του νομικού πλαισίου για το διασυνοριακό εμπόριο θα πρέπει να ενθαρρύνει και την οικονομική δραστηριότητα και να αυξάνει και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων. Οι διαφορές στους κανόνες που διέπουν το ενοχικό δίκαιο των πωλήσεων μπορεί να αποτρέψει τους ε, καταναλωτές από το να αγοράσουν και τους εμπορευόμενους από να πουλήσουν σε διασυνοριακό επίπεδο και επομένως να ε, υποσκάψει την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Ε, η πρόταση της Κομισιόν για ένα κανονισμό για ένα κοινό δίκαιο ευρωπαϊκών πωλήσεων θα δημιουργήσει ένα προαιρετικό καθεστώς για διασυνοριακές συμβάσεις για την πώληση αγαθών και την παροχή ψηφιακού περιεχομένου. Όταν επιλέξουν τα μέρη, τότε θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο και το δίκαιο αυτό θα αφορά τις, ε, τις ε, συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ή και επιχειρήσεων ειδικά όταν ένα από τα δύο μέρη είναι ΜΜΕ. Ε, το κοινό αυτό δίκαιο πολίσεων δεν θα αντικαταστήσει τους, ε, τα εθνικά δίκαια, αλλά θα λειτουργεί παράλληλα, θέλει να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασία των καταναλωτών και η πρόταση για ένα κανονισμό ενός κοινού δικαίου ευρωπαϊκών πωλήσεων είναι σημαντικό για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και το εμπόριο στην εσωτερική αγορά ε, επί τη βάση της ελευθερίας των συμβάσεων και να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Για να προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία ε, έχουμε προβλέψει έξι ημέρες συνεδριάσεων στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Και ξέρω ότι μέχρι σήμερα εξετάστηκαν όλα τα άρθρα στο, στην ομάδα του Συμβουλίου. Επίσης, ε, ξέρω ότι αυτό το μέτρο δεν έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις ε, στο Συμβούλιο. Ξέρω ότι συνεχίζονται συζητήσεις και μπορεί να επιτευχθεί συμβιβασμό που θα διευκολύνει μια ενιαία προσέγγιση μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και θα επιτρέψει σε αυτό το μέτρο, τουλάχιστον εν μέρη, να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς περαιτέρω περιτές καθυστερήσεις. Θα έχω και, και επίσημες πληροφορίες για την τύχη αυτού του κειμένου, αλλά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία στις α, επιγραμμικές συναλλαγές για το ψηφιακό περιεχόμενο. Ξέρουμε ότι για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και διασυνοριακά. Θα πρέπει λοιπόν οι καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο, ε, αλλά γι' αυτό, για να μπορούν να το κάνουν, θα πρέπει να κατανοούν καλύτερα τι προστασία τους παρέχεται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις ε, συναλλαγές στο διαδίκτυο. Ελπίζω να υπάρξει πρόοδος κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας. Ξέρω ότι υπήρξαν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, ξέρω ότι υπήρξαν διαφωνίες, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ενιαία άποψη, ούτω ώστε να έχουμε τουλάχιστον πρόοδο στις, ε, στα θέματα των επιγραμμικών συναλλαγών και να αυξήσουμε έτσι την, ε, το διασυνοριακό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή σας δεν έχει τη βασική ευθύνη για αυτή την πρόταση, το ξέρω, αλλά θέλω να πω δύο λόγια παρόλα αυτά για τον προτινόμενο κανονισμό για την προστασία των ε, δεδομένων που συνιστά μια σημαντική επικαιροποίηση τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων αυτών. Ο προτινόμενο κανονισμό έχει σαν σκοπό να αυξήσει τον έλεγχο των ατόμων ε, στα προσωπικά του δεδομένα και θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη ε, στην ψηφιακή οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε υψηλότερα επίπεδα καινοτομία, οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση. Ο κανονισμό έχει σαν σκοπό να εξασφαλίσει πιο εναρμονισμένο και απλό τρόπο εφαρμογή των προτύπων προστασία των δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξάνοντας το επίπεδο διασυνοριακής ε, δραστηριότητα στην ε, εσωτερική αγορά. Εκτιμάται ότι η αξία της ευρωπαϊκής ε, οικονομίας στο ίντερνετ στην ενιαία αγορά μπορεί να φτάσει στο 5% του ΑΕΠ τα επόμενα, του ΑΕΚ, τα επόμενα χρόνια με, και να δημιουργήσει μέχρι και 4 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση, αν εφαρμοστεί το ψηφιακό θεματολόγιο. Ο προτινόμενος κανονισμός αναγνωρίζει ότι όπως μεταφέρονται τα δεδομένα σε όλο τον κόσμο, ε, αυτό μπορεί να αυξήσει και την ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τόπου α, επιχειρηματικής δραστηριότητας και επενδυτικής δραστηριότητας. Είναι σημαντικό λοιπόν ο κανονισμός αυτός να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και ένα πιο απλό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η πρόοδος σε αυτό το μέτρο πιστεύουμε ότι θα υποστηρίξει με άμεσο τρόπο την επιχειρηματική δραστηριότητα και την ανάπτυξη. Και η πρόθεση αυτού του πακέτου είναι επίση μία από τι προτεραιότητε ε, τη προεδρία μα ε, στον τομέα τη δικαιοσύνη. Έχουν γίνει ήδη οι συνεδριάσεις στην ομάδα εργασία και υπάρχει μια θετική στάση για να σημειωθεί η πρόοδος σε αυτό το σημαντικό θέμα. Έχουμε 15 ημέρε ε, συνεδριάσεων κατά τη διάρκεια τη Ιλλανδικής Προεδρία για αυτό το σημείο. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό επίση. Δεν θέλω να κλείσω την παρουσίασή μου χωρί να πω δύο λόγια για άλλα μέτρα τα οποία ελπίζουμε ότι θα διευκολύνουν την πρόοδο και ελπίζουμε ότι θα διευκολύνουμε την πρόοδο, κάποια από αυτά τα συζητήσετε σήμερα. Δίνω ιδιαίτερη σημασία στην Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας για αστικά θέματα που θα συζητήσετε αργότερα. Είναι σημαντικό τα άτομα τα οποία ήταν θύματα, ε, ας πούμε, οικιακής βίας ε, σε ένα κράτος να έχουν μια τέτοια εντολή ε, προστασίας. Ακόμα και όταν ε, επισκέπτονται ένα άλλο κράτος μέλος, είτε για διακοπές, είτε για να διαμείνουν εκεί, δεν θα πρέπει ο βίαιος συντροφός τους να τους ακολουθήσει και να αγνοήσει την προστασία που τους δόθηκε στο πρώτο κράτος μέλος και να εκφοβήσει το άτομο αυτό, το οποίο έχει αποφεληθεί από μια τέτοια εντολή προστασίας. Είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το μέτρο. Ασχολήθηκα επί πολλά χρόνια με το οικογενειακό δίκαιο και φυσικά με ενδιαφέρει τα μάλα αυτό ο κανονισμός του Συμβουλίου για, το, για τη δικαιοδοσία, το εκτελεστέο δίκαιο και την εφαρμογή των αποφάσεων σε ό,τι αφορά το γαμικό δίκαιο και τις, συνέπειε για την περιουσία των, συντρόφων ή συζύγων. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει για αυτό το θέμα, για το τι γίνεται με την περιουσία, και αν αφορά μόνο τα κίνητα ή ας πούμε αν αφορά και τις συντάξεις και πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία. Ξέρω ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, δυσκολίσει ειδικά με τις επίσημες καταχωρημένες ε, σχέσεις. Ε, νομίζω ότι τα δύο κείμενα θα πρέπει να προωθηθούν παράλληλα. Δηλαδή αυτό για τους συζύγους και αυτό για τους επίσημους συντρόφους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε με επικοδομητικό τρόπο αυτά τα δύο θέματα. Εν κατακλείδη, η Προεδρία μας έχει μια πολύ απαιτητική ατζέντα στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης και θα προσπαθήσουμε να την εντάξουμε στις σημαντικές προτεραιότητες για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, πρόθεσης της ανάκαμψης και της δημιουργίας θέσεων απασχόληση. Είναι αμφισβήτητο ότι τα μέτρα αστικής δικαιοσύνης μπορούν να συνεισφέρουν για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να βοηθήσουν την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε στην ε, οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτά θα τα κάνουμε χωρίς να αγνοήσουμε όμως τα κοινωνικά θέματα τα οποία είναι σημαντικά ε, στον τομέα του αστικού δικαίου. Θα ήθελα τέλος να σας πω ότι ξέρω πολύ καλά ότι η δουλειά που κάνουμε και η δουλειά που κάνετε έχει άμεση επίπτωση στη ζωή εκατομμύριων Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες με επικοδομητικό τρόπο και ελπίζω να φτάσουμε τέλη Ιουνίου με ένα πακέτο μέτρων που έχουμε προωθήσει και ελπίζω αυτό να είναι υποφελές για όλους μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, κύριε Σάτερ. Πολύ περιεκτική παρουσίαση και πολύ ενδιαφέρουσα ε, για τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορώ να σας διαβεβαιώσω για την διάθεσή μας ε, για επικοδομητική συνεργασία και συνεχή ανταλλαγή απόψεων ε, μαζί σας τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά. Περνάμε τώρα Αγαπητοί συνάδελφοι, στο πρώτο μέρος ε, του εργαστηρίου μελέτης συνολικά έχουμε τρία μέρη, μην ξεχνάτε. Στο πρώτο μέρος ασχοληθούμε γενικά με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Έχουμε ήδη μια ελαφρά καθυστέρηση σε σχέση με το χρονοδιάγραμμά μας. Θα πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε πια, λίγο πιο αυστηροί με την τήρηση του χρόνου και να φροντίσουμε να μην τον ξεπερνάμε για να προλάβουμε να έχουμε και μια συζήτηση μετά την παρουσίαση των ομιλιών και ανταλλαγή απόψεων. Στις ε, εργασίες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων είχα και προσωπικά την ευκαιρία ω εισηγητής να ασχοληθώ με το θέμα της ε, κοινοτικής ενωσιακής ομοθεσίας μάλλον για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Είχαμε καταρχήν τον κανονισμό Ρώμη 3 για τα διαζύγια και τους δικαστικούς χωρισμούς με κάποιο διασυνοριακό στοιχείο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εργασία αυτή και από δικονομική και από ουσιαστική άποψη. Γιατί για πρώτη φορά έχουμε τέτοιου είδους ε, ε, νομοθεσία στην οποία εφαρμόζεται η διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας με 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφάσισαν να συσφίξουν ε, τις σχέσεις και τις συνεργασίες τους σε θέματα διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού μεταξύ συζύγων διαφορετικών ε, εθνικοτήτων ή διαφορετικών υπηκοτήτων. Και μάλιστα οι εργασίες αυτές που κάναμε έδειξαν ε, την, το μεγάλο φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλές φορές οι πολίτες που ασκούν το δικαίωμά τους ελεύθερης διακίνησης και αλλάζουν ε, την χώρα διαμονής τους ή τη χώρα εργασίας τους. Είχαμε δυσκολίες στην αναζήτηση του ελάχιστου κοινού παρανομαστή που θα είναι ικανοποιητικός και ε, ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ε, εθνικών νομοθεσιών. Ήταν τιτάνιο έργο και παρόμοια περίπτωση είχαμε και στην αναδιατύπωση ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 1. Μας τον έφερε ο καθηγητής Λέναρς, δεν πρόκειται να επανέλθω σε αυτό. Είχαμε μια πραγματικά ε, δύσκολη περίοδο, μια διετή ε, προσπάθεια και έντονες εργασίες για να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά που δεν κάλυπταν μόνο τους επιχειρηματίες αλλά και τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Το ίδιο ισχύει και για το πτωχευτικό δίκαιο. Ε, συγγνώμη, για το κληρονομικό δίκαιο. Είχαμε σημαντικά θέματα γιατί υπήρχαν αρκετά κενά και τεράστια νομικά κολλήματα αλλά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν ε, οι πολίτες και μάλιστα σε μια δύσκολη κατάσταση της ζωής όταν ε, έχαναν κάποιο συγκινικό τους ε, κοντινό τους άνθρωπο και ταυτόχρονα είχαν να αντιμετωπίσουν τα κενά στο κληρονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ε, υπήρχαν προβλήματα και στις εμπορικές συναλλαγές με όλο και μεγαλύτερη κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Η διευρυμένες αυτές οι εμπορικές συναλλαγές και η ενισχυμένη ελεύθερη διακίνηση δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προβλήματα. Γιατί αναδεικνύεται η ανάγκη μεγαλύτερης ενοποίησης, εναρμόνισης των νομικών διατάξεων για να έχουμε δυνατότητα για ταχύτερη αλλά και ευθυνότερη επίλυση των προβλημάτων και των συμπολιτών μας αλλά και των επιχειρηματών των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων που προσκούρουν μερικές φορές στις διαφορετικές διατάξεις ε, του δικαίου και προκειμένου του αστικού δικαίου. Ε, υπάρχει το θέμα της αυτόματης αναγνώρισης των ε, δικαστικών αποφάσεων ή κάποιων ε, πράξεων αστικού χαρακτήρα, κάτι που ενισχύει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαιικών συστημάτων και μάλιστα αυτό οφείλεται και στην ενίσχυση της διακίνησης, αλλά και στην εξοικείωση με τα διάφορα συστήματα δικαίου. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με όλα, αυτά τα θέματα, ε, για τα οποία χρειαζόμαστε κοινέ διατάξεις ε, κοινοτικέ χάρη των Ευρωπαίων πολιτών. Και όλες οι νέες ε, νομοθετικές προτάσεις είναι απόρρια των καταστάσεων που δημιουργούνται και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτε μα στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά και στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησής τους. Ε, εξετάστηκε και η πρόταση για ένα ευρωπαϊκό κώδικα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, η εναρμόνιση κάποιων διατάξεων ε, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Όλες αυτές είναι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μεταξύ άλλων και στη σημερινή μας συνεδρία, στο σημερινό μας εργαστήριο μελέτης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Παρασκευή Μίσου που είναι ε, Διευθύντρια της Αστικής Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you, Chair. Honor... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τιμή και χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτό το εργαστήριο μελέτης. Είναι μια ουσιώδη συζήτηση, ούτως ώστε το 2013 να είναι ένα ευτυχές έτος για τους πολίτες. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό? Σήμερα ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δικαιοσύνης είναι απτή πραγματικότητα. Τόσο απτή όσο η ενιαία αγορά και η ΟΝΕ η δικαιοσύνη, η ηθαγένεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι αξίες κλειδιά. Ουσιώδες τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Οι πολίτες μπορούν να ασκήσουν ουσιοδός τα δικαιώματά τους, ταξιδεύοντας, μετακινούμενοι προσωρινά ή μόνιμα σε μια άλλη χώρα της Ένωσης για να σπουδάσουν, να εργαστούν να ξεκινήσουν μια οικογένεια, μια επιχείρηση ή να συνταξιοδοτηθούν. Έχει επιτευχθεί πρόοδος στο αστικό και εμπορικό δίκαιο και οι σχέσεις με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο έχουν περαιτέρω δημιουργηθεί. Οι πολίτες τώρα έχουν ε, απλούστερα και ταχύτερα κανάλια για να επιβάλλουν τα αιτήματά τους σε διασυνοριακά θέματα ιδίως μετά την εφαρμογή της ε, Σύμβασης Βρυξέλλες 1, όπου εσείς ήσασταν εισηγητής. Από το 2015 θα υπάρχει δυνατότητα επιβολής δικαίου γενικώ στην Ένωση. Οι πολίτες εποφελούνται από ισχυρότερα δικαιώματα ως καταναλωτές κατά τις επιγραμμικές συναλλαγές και υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε κοινού κανόνες για θέματα ε, αστικής υπετότητας και συμβολέων. Η προστασία των ε, γυναικών και των συζύγων έχει βελτιωθεί, ούτω ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι μετά από ένα χωρισμό τα παιδιά μπορούν να διατηρήσουν τακτική ε, επαφή με τους γονείς τους και η επιμέλειά τους χρηματοδοτείται. Αύριο θα έχουμε κανόνες για όλες τις πλευρές της ζωής των πολιτών. Για την κληρονομία και για τα διαζύγια έχουμε δύο κανονισμούς που έχουν εγκριθεί για τα περιουσιακά στοιχεία των συζύγων. Έχουμε δύο προτάσεις υποσυζήτηση και θα υπάρξει και για τα δημόσια έγγραφα μία πρωτοβουλία. Ούτω ώστε να διευκολύνουμε περαιτέρω τη ζωή των πολιτών όταν μετακινούνται στο εξωτερικό. Επίσης ε, εργαζόμεθα για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Πολίσεων, όπως είπε και ο Υπουργός. Αυτό είναι ιδιαίτερα χάρη και στους εισηγητές κυρίους Λένε και Μπερλίνγκουερ. Στα πρόθυρα της έναρξης του 2013 ως έτους ε, των πολιτών, η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ είπε ότι οι πολίτες θέλουν συγκεκριμένα αποτελέσματα από την Ευρώπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Η αστική δικαιοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων. Και μεταξύ των ε, διαθέσιμων λύσεων πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία του δικαστικού τομέα και να προωθήσουμε την δικαιοσύνη για την ανάπτυξη. Σε αυτό το σημείο των αναζητήσεών μας η Επιτροπή είναι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι έκανε μια αναλυτική μελέτη για το ευρωπαϊκό πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ε, τα, ε, τις ελλείψεις και τις περαιτέρω προοπτικές. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Κομισιόν θα προτείνουμε νέα νομοθετήματα για να κλείσουμε τα κενά σε αυτό το τομέα και για να υπάρξει μια κωδικοποίηση του αστικού κεκτημένου. Έχουμε συνέστηση της ε, ευθύνης μας για να ολοκληρώσουμε για τα αστικά θέματα τη δικαιοσύνη και θα ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη που δημιουργήθηκε για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκόλμης. Φέτος, αλλά και του χρόνου, θα προτείνουμε και θα συμβάλλουμε περαιτέρω στην εργασία σε αυτόν τον τομέα. Αλλά παράλληλα, ενθαρρύνουμε τις έρευνες και συζητήσεις έχοντας υπόψη όμως ότι οι προτάσεις για κωδικοποίηση είναι σημείο κίνησης της πολιτικής συζήτησης ε, στον τομέα αυτό. Οπότε σημαντικές προκλήσεις και ερωτήσεις πρέπει να τύχουν απάντησης πριν ξεκινήσουμε. Πολύ σύντομα να αναφερθώ σε μερικά μέτρα της ε, δικαιοσύνης για την ανάπτυξη όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά και από τον Υπουργό. Πρώτον, προτάσεις για την εγκυότητα. Τις εγκρίναμε. Τις υποβάλαμε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 12 Δεκάτου. Και επίσης υπήρξε και μια ανακοίνωση. Ο κύριος Υπουργός μας είπε τι περιλαμβάνει ο κανονισμός. Πολύ Καλά, αλλά είναι μόνο ένα πρώτο βήμα, θέλω να τονίσω αυτός ο κανονισμός. Μετά την ανακοίνωση που επίσης ενέκρινε η Επιτροπή, θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία συζήτησης για ε, μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την αποτυχία των επιχειρήσεων και την πτώχευση. Θέλουμε να κάνουμε μια δημόσια διαβούλευση, ούτω ώστε να υπάρξει μια κουλτούρα διάσωση και αναδιάρθρωσης, ανάκαμψη των επιχειρήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν οικονομικά δυσχερείς καταστάσεις. Για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες που ε, πτωχεύουν τιμίως θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μια, από μια περίοδο να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. Η Επιτροπή ε, ελπίζει να τύχει υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε το θέμα αυτό να λάβει την αναγκαία προτεραιότητα και σημασία. Και επίσης υπάρχει και η πρόταση για μια διαταγή, ευρωπαϊκή διαταγή διατήρηση λογαριασμού, όπου ο εισηγητής κ. Μπαλτασάρε έχει σημειώσει πρόοδο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καταλήγω. Υπάρχουν μια σειρά άλλες προτάσεις που ανέφερε ο υπουργό, αλλά καταλήγοντας λέω ότι προσβλέπω σε ταχεία πρόοδο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο επί αυτών αλλά και επί του ε, συμβατικού δικαίου κατά την Ιρλανδική Προεδρία. Πρόκειται για την 7η Ιρλανδική Προεδρία και πιστεύω ότι θα καθοδηγήσουν επιτυχέστατα τη διαδικασία αυτή. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για την Προεδρία τους, ούτως ώστε να εγκριθούν αυτά τα μέτρα που θα προσδώσουν περισσότερη ασφάλεια δικαίου, θα συμβάλλουν λοιπόν στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, θα ωφελήσουν τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μίχου. Το επόμενο θέμα είναι η οδηγία για ορισμένα θέματα της διαμεσολάβησης στον αστικό και εμπορικό τομέα δύο μιλητές. Πρώτος, ο συνάδελφός μου, η συνάδελφός μου, Άλεν Μακάρτη, τη Νομική Επιτροπή. Ευχαριστώ χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω την εργασία που κάνουμε στην Νομική Επιτροπή και που υποστηρίζεται και έχει επικυρωθεί από ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Καταρχάς, ως πολιτικός, ως νομοθέτης λαμβάνω αιτήματα βοήθειας από τους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας που πολλές φορές αφορούν διασυνοριακά θέματα, θέματα επιμέλειας, δαιμονίας, πρόσβαση στα παιδιά, ε, διατροφή, ιδιοκτησιακά θέματα, θέματα επιχειρήσεων Έρχονται λοιπόν σε εμά ω εκπροσώπου των για να του βοηθήσουμε να επιλύσουν τα θέματα αυτά. Και από τι υποθέσει που με απασχολούν, ξέρουμε ότι οι αντιδικίε στο δικαστήριο είναι δαπανηρέ. Σε μία μελέτη, 45% των πολιτών που ερωτήθηκαν είπαν ότι δεν θα προσέφεραν σε δικαστήρια άλλης χώρας εάν το αμφισβητούμενο ποσό είναι λιγότερο από 50.000 ευρώ γιατί φοβούνται ότι θα πλήρωναν περισσότερο σε δικαστικά έξοδα. Όλα αυτά τα ευρήματα μας αποδεικνύουν ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι πολύ πολύτιμο εργαλείο για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις. Αυτό θέλουμε να πούμε στα κράτη-μέλη. Πρέπει να κάνουν περισσότερο για να προωθήσουν τα ωφέλη της διαμεσολάβησης, της διαιτησίας να υπάρχει για παράδειγμα κατάρτιση των ε, διαμεσολαβητών και η έρευνα μας έδειξε ότι οι βέλτιστες πρακτικές στην ε, διαμεσολάβηση οδηγούν σε 70% επιτυχία που φτάνει ως και το 80% εάν έχουν επιλέξει εθελουσίως ε, οι αντίδικοι την διαμεσολάβηση και μόνο 1% αυτή τη στιγμή όμω ε, αυτών που έχουν διαφορέ στρέφονται στη διαμεσολάβηση. Να λοιπόν ένα τεράστιο κενό μεταξύ του πόσο ωφέλιμη είναι η διαμεσολάβηση και πόσο λίγοι απευθύνονται σε αυτή. Έτσι μέσω τη διαμεσολάβηση κερδίζουμε χρόνο, κερδίζουμε χρήματα, διότι να περάσουμε στο δικαστήριο μπορεί να ε, σημαίνει 300, 300 περισσότερες μέρες και πολύ περισσότερα χρήματα. Και από το κράτο μέλο από όπου προέρχομαι ξέρουμε ότι η αντιδικία πολλές φορές ως μέσο όρο καλύτερα διαρκεί 333 μέρες και κοστίζει 35.000 ευρώ ενώ ε, εάν είχαν ε, περάσει στη διαμεσολάβηση θα είχε διαρκέσει κατά μέσο 35 μέρες και θα κόστιζε πολύ λιγότερα. Σαφή λοιπόν τα ωφέλη. Ένας διαμεσολαβητής μου είπε ότι ε, μέσα σε ένα χρόνο αντιμετώπισε 150 υποθέσεις, οι 100 από αυτές επιλήθηκαν σε μια εβδομάδα. Εδώ στο Βέλγιο υπάρχουν χίλιοι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και ε, υπάρχουν 600.000 υποθέσεις στα δικαστήρια ενώ πολύ λιγότερες περνάνε στη διαμεσολάβηση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αυτή η οδηγία, πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ένωση. Εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2008 μετά από συμφωνία με το Συμβούλιο Είχαμε δύο επιτυχείς ακροάσεις προηγουμένως το 2006 το 2007 και επίσης είχαμε και μια επιγραμμική διαβούλευση. Πρώτη φορά που η Επιτροπή μας αποφάσισε να κάνει τέτοιου τύπου διαβούλευση για να υπάρξουν πολλές συμμετοχέ από όλες τις χώρες της Ένωσης. Και τι είδαμε σε αυτήν την ε, διαβούλευση και μας έπεισε μάλιστα ήταν ότι η οδηγία εκείνη τη στιγμή για την οποία ε, πολλοί είχαν επιφυλάξει, ήταν πολύ καλή ιδέα γιατί είδαμε πόσο η κοινή γνώμη ήθελε να υπάρξει μια τέτοια οδηγία. Αυτή η οδηγία διευκολύνει τη διαμεσολάβηση, ενισχύει τι νομικέ εγγυήσει που τη συνοδεύουν και πιστεύουμε ότι αυτό βοηθάει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις. Κάθε δικαστής έχει τη δυνατότητα να προτείνει να ε, παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι μια ενημέρωση για τη διαμεσολάβηση και εάν συμφωνήσουν να προτείνουν τη διαμεσολάβηση. Έτσι οι διάδικοι μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία η οποία έχει περίπου το, ε, την ίδια νομική αξία με μια δικαστική απόφαση που μετά μπορεί να εγκριθεί και να περάσει και από συμβολιογράφου και μπορεί να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη με τι υπάρχουσε νομικέ ρυθμίσει. Η οδηγία αυτή διασφαλίζει ότι η διαμεσολάβηση πρέπει να γίνει σε ατμόσφαιρα εμπιστευτικότητα. Και η πληροφορία που ε, ε, δίδεται, οι καταθέσει δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά των ε, εμπλεκομένων σε ε, ένδικες διαδικασίες αργότερα αν αποτύχει διαμεσολάβηση. Αυτό είναι ουσιώδες για να υπάρχει αναγκαία εμπιστοσύνη, για να ε, ενθαρρύνουμε την χρήση της διαμεσολάβησης. Γι' αυτό η οδηγία προβλέπει ότι δεν είναι δυνατόν να ε, οι εμπλεκόμενοι να υποχρεωθούν να ενημερώσουν για το τι έγινε κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. Και επίσης για τις περιόδους παραγραφής και περιορισμού υπάρχουν οι αναγκαίες διατάξεις ούτως ώστε να αναβάλλεται όταν υπάρχει διαμεσολάβηση, να αναστέλλεται μάλλον όταν υπάρχει διαμεσολάβηση ή η προθεσμία παραγραφή ούτω ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα να προσφύγουν αργότερα στη δικαιοσύνη. Έτσι διατηρείται το δικαίωμα προσφυγή στη δικαιοσύνη αν αποτύχει μεσολάβηση. Όσο πλησίαζε η προθεσμία για την έναρξη εφαρμογή, αποφασίσαμε να κάνουμε μία έκθεση για την εφαρμογή τη διαμεσολάβηση. Η Δανία, όπω ξέρετε, δεν συμμετέχει σε διαμεσολάβηση, ενώ η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν να συμμετάσχουν. Δεν μπορώ να σα αναλύσω τώρα πώ έχει εφαρμοστεί αναλυτικά αυτή η οδηγία, αλλά αναφέρω ορισμένα στοιχεία που νομίζω ότι ενδιαφέρουν για το πώ εφαρμόζεται στα διάφορα κράτη-μέλη. Το άρθρο 1.2 αναφέρει ότι η οδηγία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε διασυνοριακέ υποθέσει. Εδώ υπήρξε μάχη μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχασε Διαπιστώσαμε όμως ότι οι περισσότερες εθνικές νομοθεσίες δεν κάνουν τη διάκριση μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών ε, προστριβών, οπότε στην ουσία εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο. Για την εγγύηση εμπιστευτικότητα, στο άρθρο 7, τα περισσότερα κράτη-μέλη την εγγυούνται και προστατεύουν ε, τους συμμετέχοντες από το να είναι υποχρεωμένοι να ε, καταθέσουν για το τι έγινε. Στην Ιταλία το άρθρο 10 του δικού τους νομοθετικού διατάγματος λέει ότι όσα γίνονται, όσα λέγονται κατά τη διαμεσολάβηση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω δικαστικές ένδικες διαδικασίες. Και το άρθρο 9 λέει ότι οποιοδήποτε συμμετέχει στη διαδικασία διαμεσολάβησης έχει υποχρέωση εμπιστευτικότητα. Για οτιδήποτε έχει υποθεί ή όποια πληροφορία έχει κατατεθεί κατά τη διάρκεια τη διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να ε, θεωρήσει και να τηρήσει την πληροφόρηση εμπιστευτική εκτός αν ε, οι ε, εμπλεκόμενοι συμφωνήσουν. Και το ίδιο ισχύει και στη Γερμανία. Και δίνει στη διαμεσολαβητή στη Γερμανία το δικαίωμα να αρνηθεί να δώσει, να καταθέσει σε ένδικες διαδικασίες για το τι υπόθηκε. Στη Σουηδία όμως φαίνεται ότι οι υποχρεώσεις είναι διαφορετικές για την οδηγία αυτή. Διότι στο άρθρο 3 των κανόνων του ε, επιμελητηρίου, του εμπορικού επιμελητηρίου, λέγεται ότι δεν είναι υποχρεωτική εμπιστευτικότητα, ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι εμπλεκόμενοι σε αυτό. Το άρθρο 3 υποχρεώνει όλους τους εμπλεκόμενους και τον διαμεσολαβητή να σεβαστεί την εμπιστευτικότητα, αλλά δεν απαγορεύει την, ε, ε, το ενδεχόμενο ο μεσολαβητής να καταθέσει ως μάρτυρα στο δικαστήριο αργότερα στις περισσότερες χώρες μέλη, τα κράτη-μέλη έχουν διαδικασία ούτω ώστε η απόφαση της διαμεσολάβησης να έχει το ίδιο καθεστώς με δικαστική απόφαση. Αυτό γίνεται είτε μέσω υποβολής της στο δικαστήριο, είτε μέσω επικύρωσής της. Στην ε, Ελλάδα το άρθρο 9 του νόμου 398 λέει ότι το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης ε, ε, υποβάλλεται μαζί με τα πρακτικά που έχουν υπογράψει οι διάδικοι και οι ε, δικηγόροι τους στα πρωτοβάθμια δικαστήρια και κατόπιν είναι εκτελεστέο. Το ίδιο ισχύει και στη Σλοβενία, όπου πρέπει να περάσουν από συμβολιογράφων. Το άλλο θέμα για μας όσον αφορά την παραγραφή Ε, όπου λοιπόν έχει, προβλέπεται παραγραφή έχει καθοριστεί ότι δεν πρέπει η διαμεσολάβηση να περιορίζει τη δυνατότητα περαιτέρω προσφυγής στα δικαστήρια διότι αναστέλλεται η ε, προθεσμία λοιπόν για παραγραφή. Σε άλλες χώρες έχουν πάει περισσότερο, έχουν πάει πιο μακριά και ε, πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη περισσότερο η διαμεσολάβηση. Και γι' αυτό η διαμεσολάβηση ε, είναι αντικείμενο κινήτρων. Χορηγεί το κράτος κίνητρα. Για παράδειγμα, ε, λαμβάνουν κάποια επιστροφή των ε, εξόδων τους εάν επιληθεί επιτυχώς μέσω διαμεσολάβησης. Στη Βουλγαρία λαμβάνουν το 50%, στη Ρουμανία το 100% του κόστους. Σε ορισμένες χώρες είναι υποχρεωτική η διαμεσολάβηση. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει πρώτα να γίνει προσπάθεια διαμεσολάβησης και μόνο μετά μπορούν να περάσουν σε ένδικη διαδικασία. Αυτό ισχύει για το οικογενειακό δίκαιο. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει για αστικά και εμπορικά θέματα οπωσδήποτε να περάσουν πρώτα από διαμεσολάβηση. Το διάταγμα 28 που άρχισε να ισχύει στις 21 Μαρτίου 2011 στοχεύει να τροποποιήσει το, νομοθετικό, το δικαστικό σύστημα και με αυτόν τον τρόπο να μειώσει ε, την καθυστέρηση εκδίκαση υποθέσεων γιατί αυτή τη στιγμή μέσω, ο μέσος όρος ε, διάρκειας μιας υπόθεσης είναι 9 χρόνια. Αυτό φυσικά δεν ικανοποίησε τους δικηγόρους, που μάλιστα απέργησαν γι' αυτό. Πολύ πρόσφατα υπήρξε προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή από πλευρά της Επιτροπής μας κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, όπου ζητήσαμε ε, να υπάρξει περισσότερη πρόοδος για τη διαμεσολάβηση και να αυξηθεί η εφαρμογή της παντού στην Ένωση. Πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα πήγον το θέμα αυτό λόγω ε, της περίοδου λιτότητας και κρίσης ε, που ε, ζούμε και γι' αυτό πρέπει να μεθεί το κόστος και ο χρόνος για την επίλυση των δικαστικών αντιφάσεων, ε, των δικαστικών υποθέσεων. Από τη μία έχουμε όλα τα στοιχεία όμως που μας λένε ότι ακόμη και αν επιτύχει περιορισμένα η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος εκδίκασης αλλά από την άλλη μεριά είναι αποκοτευτικά λίγες οι υποθέσεις που πάνε σε διαμεσολάβηση παντού στην Ένωση και αυτό ακριβώς δεν θέλαμε όταν εγκρίναμε αυτή την οδηγία ως θεσμικά όργανα. Γι' αυτό καλούμε την Επιτροπή να υπάρξει περισσότερη πρόοδος για να επιτευχθούν οι στόχοι της ε, οδηγίας ταχαίως. Καλούμε την Επιτροπή να διασφαλίσει την σωστή ισορροπία μεταξύ μεσολάβησης και ένδικων μέσων καλούμε την Επιτροπή να προσπαθήσει να επιτύχει αυτήν την ε, ε, καλύτερη εξισορρόπηση τουλάχιστον να αυξηθεί η διαμεσολάβηση σε δύο μεθεωριακές υποθέσεις και θα θέλαμε να δούμε πώς θα μας βοηθήσει η Επιτροπή να υπάρξουν μίνιμουμ ποσοστά για την επίλυση διαφορών σε ορισμένες υποθέσεις. Διάβασα τις προθέσεις της Επιτρόπου Ρέντινγκ, την πρόθεσή της να υπάρξει ανακοίνωση του χρόνου για την διαμεσολάβηση για να προωθηθεί περαιτέρω η χρήση της και από ό,τι κατάλαβα από τις προσωπικές μου επαφές με την Επίτροπο ξέρω ότι συλλέγει αναλυτική πληροφόρηση για το πώς εφαρμόζεται η οδηγία αυτή στα κράτη-μέλη. Καταλήγοντας, προσβλέπουμε στην έκθεση του 2016 που θα μας υποβληθεί από την Επιτροπή με βάση τις εθνικές εκθέσεις που έχουν ζητηθεί από τα κράτη-μέλη από την Επιτροπή εξακολουθούμε ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή, να πιστεύουμε ότι είναι ευέλικτο, ταχύ και φθηνό μέσο επίλυσης διαφορών, επιτρέπουν περισσότερο έλεγχο στους ε, αντιδίκους, ε, τους δίνει περισσότερη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών, βοηθά ιδιαίτερα σε ε, θέματα οικογενειακού δικαίου που αφορούν τα παιδιά, γιατί πολύ γρήγορα καταλήγουν σε αποφάσεις για την ευημερία των παιδιών, για την ευημερία συνολικά της οικογένειας που αντιμετωπίζει καταστάσεις άγχους και σύγκρουσης. Ευχαριστώ. Ελπίζω ε, να μου δώσετε δυνατότητα να απαντήσω σε ερωτήσεις, αλλά πρέπει να πάω κι αλλού για μια άλλη ομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μακάρθη. Ε, niezwykle ε, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ομιλία σας, ε, κυρία Μακάρθη. Είστε άλλωστε η Δήμον στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων για θέματα διαμεσολάβηση και φάνηκε αυτό από την πολύ μεστή παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε προβλέψει και γύρω ερωταπαντήσεων και μάλιστα σας έχουμε μοιράσει και έντυπο για να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχή στη συζήτηση. Η γραμματεία θα μαζέψει τα έγγραφα, τους καταλόγους. Ωραία. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Στέφεν ε, Στάουτιγκερ που μας ήρθε από τη Βιέννη δι είναι συμβολογράφος ε, και επίσης ο Δ. Πρέιερ ε, ειδικεύεται σε θέματα διαμεσολάβηση. Έχετε το λόγο. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να θέσω μία ερώτηση. Ποιος από εσά έχει παρακολουθήσει κατάρτιση διαμεσολαβητή, σεμινάριο διαμεσολαβητή. Δεύτερη ερώτηση. Ποιος από εσά έχει εμπειρία σε θέματα διαμεσολάβησης, ποιος συμμετείχε σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης και ποιος έχει μια θετική εμπειρία από μια διαμεσολάβηση. Μάλιστα. Γιατί θέμα της δικής μου ομιλία είναι γιατί η διαμεσολάβηση ως σύστημα, εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών δεν χρησιμοποιείται συχνότερα. Και μάλιστα στην ερώτηση αυτή υπονοούμε ότι η διαμεσολάβηση είναι κάτι θετικό. Είναι μια ε, εποφελής ε, διαδικασία και διαρωτώ με τι θα άλλαζε αν προσφεύγαμε πιο συχνά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια αποτελεσματική διαμεσολάβηση και πώς μπορούμε να κρίνουμε ότι είναι αποτελεσματική αυτή η διαδικασία. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχει και ένα θέμα ε, οικονομικό, μήπως ε, και υπάρχει ένας πόλεμος στην μερικές φορές που γίνεται, όταν είναι χρονοβόρη διαδικασία. Ποιο είναι το οικονομικό της τίμημα και ποια είναι τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης. Με βάση το αυστριακό δίκαιο υπάρχει μια γραπτή συμφωνία ε, διαμεσολάβησης που γίνεται εξοδικαστικά. Αλλά δεν είναι δωρεάν. Το τίμημα είναι 1% της ε, αξίας ε, του αντικειμένου της αγωγής. Δεν ξέρω αν κάποιος θεωρεί ότι είναι υπερβολικό αυτό το τίμημα για τη διαμεσολάβηση. Μία τέτοια εισφόρα ε, θεωρούν πολλοί ότι θα πρέπει να καταργηθεί, να είναι τελείως δωρεάν η διαμεσολάβηση, να μην είναι τμήμα της επίδικης αξίας. Πολύ συχνά τη βλέπουμε από το πρίσμα της μείωσης του κόστους, αλλά δεν θα πρέπει να υπερτιμούμε αυτό το επιχείρημα. Ξέρετε ότι η διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική δυνατότητα. Βεβαίως πρέπει να έχει λοιπόν ορισμένα πλεονεκτήματα. Αλλά ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Είναι η ευθύνη για τον εαυτό τους. Αυτό δίνει δυνατότητα στους ανθρώπους σε δυνατότητες σύγκρουσης να καθορίσουν οι ίδιοι την ε, ποιότητα της ζωής τους. Το ερώτημά μου είναι αυξάνει την ποιότητα της ζωής. Για να το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι έχουμε μεγάλες δυσχέρειες. Όποιος δεν έχει εμπειρία τέτοιου ε, γεγονότος δεν μπορεί να, το, να πιστεί για κάτι τέτοιο μόνο μέσω ενός άρθρου εφημερίδας ή μιας διαφήμισης εφημερίδας. Κάτι άλλο. Η σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και δικηγόρων. Η διαμεσολάβηση ε, είναι πιο φτηνή και άρα δεν χρειάζονται δικηγόροι που είναι από ό,τι λέγεται. Είναι ακριβή. Βεβαίω ε, είναι κατανοητό ότι οι δικηγόροι ε, δεν χαίρονται να ακούγονται τέτοια επιχειρήματα. Και λένε αντίθετα ότι πολλοί διαμεσολαβητές δεν είναι επαρκώς νομικώς καταρτισμένοι. Και άρα τα αποτελέσματα των διαδικασιών ε, με διαμεσολάβησης είναι πολλές φορές νομικώς αμφισβητήσιμα. Κατανοητό αυτό το επιχείρημα. Εγώ τώρα είμαι συμβολιογράφος. Οι συμβολιογράφοι είναι πεισμένοι εξορισμού, εγγενετής, ότι είναι γεννημένοι διαμεσολαβητές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όσων δεν έχουν επαρκή πείρα διαμεσολάβησης. Ε, είμαι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε αυτό. Φυσικά οι οι συμβολιογράφοι προσπαθούν πολλές φορές να διαμεσολαβήσουν. Αλλά η διαμεσολάβηση είναι κάτι διαφορετικό στην Αυστρία. Εδώ έχουμε υποχρεώσεις για τους ε, συμβολιογράφους να προσπαθούν να επιτύχουν μια συμφωνία μεταξύ ε, των ε, ε, πλευρών που έχουν κάποια διαφορά. Αυτό όμως χρειάζεται ορισμένε γνώσεις. Θα πετούσα εγώ αυτοί που έχουν πείρα ενασχόλησης με διαφορές να είναι οπωσδήποτε υποχρεωμένοι να καταρτιστούν τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Κάτι άλλο. πώς θα έχουν πρόσβαση τα μέρη, τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν με διαφορά, πώς θα έχουν πρόσβαση στην ε, διαμεσολάβηση, στον διαμεσολαβητή. Εδώ και κάποιο χρόνο στην Αυστρία έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που καλεί τα δικαστήρια να δώσουν πληροφορίες ε, στους, ε, στα, στους διαδίκους για τη διαμεσολάβηση. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η διαμεσολάβηση δεν είναι αναγνωρισμένο επάγγελμα. Ο καθένας στην Αυστρία μπορεί να ορίσει τον εαυτό του ε, διαμεσολαβητή και χωρίς άλλες προϋποθέσεις να ασκήσει αυτή την ιδιότητα. Αυτό είναι αμφισβητήσιμο. Πρέπει να υπάρξει πρώτα κατά τη γνώμη μου αρκετά εμπεριστατωμένη κατάρτιση και πρέπει να υπάρχει και ασφάλιση, ασφαλιστική προστασία. Το κεντρικό πρόβλημα ωστόσο για μένα είναι ότι οι διάδικοι πολλές φορές δεν είναι διαδεθειμένοι να βοηθήσουν να επιτύχει η διαμεσολάβηση. Η εθελούσια προσφυγή είναι προϋπόθεση. Να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους επίσης οι, οι άνθρωποι που προσφεύγουν στη διαμεσολάβηση. Και επίσης εμπιστευτικότητα. Εμπιστευτικότητα σημαίνει και εμπιστοσύνη. Πολλές φορές οι προσφεύγοντες στην ε, διαμεσολάβηση δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήδη οι νέοι στο σχολείο θα πρέπει να ενημερώνονται για ηθικά θέματα, να ενημερώνονται για τους βασικούς κανόνες της ενημέρωσης. Στο σχολείο λοιπόν πρέπει να υπάρχουν θέματα ηθικής κατάρτισης. Να μάθουν οι νέοι να εκτιμούν τους άλλους και να φέρονται με εκτίμηση προς τους άλλους. Νομίζω ότι ανέφερα έτσι κάποια προβλήματα μόνο. Να σε ενημερώσω τώρα για τα τελευταία σχόλια για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης που έχει εκδοθεί πέρυσι στη Γερμανία. Μια φράση μόνο η διαμεσολάβηση Πρέπει πέρα από την επίλυση της συγκεκριμένης σύγκρουσης να συμβάλλει οι συμμετέχοντες να εκπαιδεύονται για το πώς στον τρόπο, στο μέλλον θα μπορούν με καλύτερη επικοινωνία να αντιμετωπίζουν μόνοι τα προβλήματά τους και όχι να στρέφονται ταχαίως σε τρίτους για την επίλυση των διαφορών τους. Εάν λειτουργεί η διαμεσολάβηση, έχει επιπτώσεις ευρύτερα στην κοινωνία. Εάν μέσω της διαμεσολάβησης αποκτούν ικανότητες οι άνθρωποι που θα τους βοηθήσουν κατόπιν να επιλύσουν περαιτέρω προβλήματα, τότε, μακροπρόθεσμα, θα επιτύχουμε να λύνουν μόνοι τους τις διαφορές τους. Και αυτή είναι ο στόχος που πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Δόκτωρα Πρέιερ. Επιστρέφουμε τώρα στο προηγούμενο τμήμα, στην προηγούμενη ενότητα του πρώτου μέρους. Χρειάστηκε να αντιστρέψουμε τη σειρά των θεμάτων εξαιτίας ανηλυμένης υποχρέωσης της κυρίας Μακάρθη που δεν μπορούσε να λάβει το λόγο αργότερα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην καθηγήτρια Σάντρα Κράμερ από το Τμήμα Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Εράσμους του Ρότερνταμ. Η κυρία Κράμερ θα μας παρουσιάσει τη μελέτη με θέμα τα κενά και τις μελλοντικές προοπτικές ενός Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Έχετε το λόγο. Κυρία Κράμερ. Thank you. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μετά την παρουσίαση της μελέτης ε, που σας έκανα το Δεκέμβριο, σήμερα δεν θα μιλήσω Ολλανδικά όπως την προηγούμενη φορά, αλλά Αγγλικά. Ευχαριστώ λοιπόν το Κοινοβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερος για την ανάμειξή του στο σημαντικό ζήτημα του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου και είναι πολύ ποιοτική η, εισφορά, η συνεισφορά, η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακούσαμε και τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας και ακούσαμε και την ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, όλα αυτά βαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, το, το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο εφαρμόζεται όταν μια νομική σχέση έχει ένα διασυνοριακό στοιχείο. Και από αυτή την άποψη είναι τμήμα με βάση τη γνώμη μερικών του ιδιωτικού δικαίου. Βέβαια, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο κατά παράδοση ήταν αρμοδιότητα του εθνικού δικαίου. Ο εθνικός νομοθέτης ρυθμίζει αυτά τα θέματα και σε κάποιο βαθμό καλύπτεται και από τις διεθνείς συνθήκες, όπως η Σύμβαση της Χάγης για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο από, τις ε, διευρυμένες, από τότε που κατοχυρώθηκαν διευρυμένες προεδρίες ε, της, ε, συνθήκης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997, ενεπλάκησε η διαδικασία αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργήθηκε ένα ευρύ πλέγμα κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Δεν είναι πλήρως όμως αυτό το πλέγμα, εξού και η μελέτη που καταρτήσαμε και που ο στόχο είχε να εντοπίσει τα κενά που υπάρχουν στο ε, κοινοτικό πλαίσιο του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου να εξετάσει πού χρειάζεται συμπλήρωμα αυτό το πλέγμα και επίσης να δώσει μια απάντηση στην ερώτηση του κατά πόσο ένα πιο περιεκτικό πλαίσιο ή ένα γνήσιο, ένα ουσιαστικό ευρωπαϊκό διεθνές ιδιωτικό δίκαιο απαιτείται και μάλιστα με ποιο τρόπο μπορούμε να το θεσπίσουμε. Η σημερινή μου ομιλία θα επικεντρωθεί στα τρία βασικά θέματα ΔΙΔ, την διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων. Θα επικεντρωθώ σε αυτά και θέματα ενδιαφέροντα όπως ε, η διαμεσολάβηση, η δέσμευση ε, τραπεζικών λογαριασμών μένουν εκτός ε, της σημερινής μου ομιλίας, γιατί δεν προλαβαίνω να τα καλύψω όλα. Τι σχέση έχουν λοιπόν οι κανόνε διεθνούς δικαίου, οι κανόνε διεθνού δικαδοσίας, συγγνώμη, για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά συμβάλλει στη εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και στην ε, υλοποίηση τη ελεύθερη διακίνηση. Οι κανόνε του διεθνούς συνθετικού δικαίου θα αυξήσουν τη διαφάνεια των κανόνων που διέπουν τι διασυνοριακέ σχέσει, είτε αφορούν αυτέ οικογενειακό δίκαιο, είτε εμπορικό δίκαιο, εμπορικέ συναλλαγές, και επίσης ε, την περίπτωση που οι καταναλωτές θέλουν να αγοράσουν αγαθά είτε μέσω του διαδικτύου είτε σε άλλη χώρα από αυτή τη διαμονή του. Αυτοί οι κανόνε είναι πολύ σημαντικοί για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, γιατί μια γνήσια ευρωπαϊκή ηθαγένεια και η αρχή τη ε, μη διακριτική μεταχείριση μπορεί να ελοποιηθούν μόνο εφόσον εξασφαλίζεται ίση ισότιμη μεταχείριση σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Είναι αυτονόητο ότι ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων διεθνούς ιδιωτικού δικαίου θα ωφελήσει και τα εθνικά μας δικαστήρια και τους όσους καλούνται να εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες. Τώρα, για το υπάρχον πλαίσιο. Αναλύσαμε στη μελέτη το υπάρχον πλαίσιο και διαπιστώσαμε ότι στα πλαίσια του άρθρου 81 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονται εκτεταμένες αρμοδιότητες. Οι κανόνες διεθνούς ιδιωτικού δικαίου καλύπτουν ε, πολλές κανόνες ε, ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου. Με εξαίρεση το οικογενειακό δίκαιο για το οποίο απαιτείται ομοφωνία, κάτι που ε, καθιστά πιο δύσκολη τη θέσπιση νομοθεσίας στον τομέα αυτό, όπως έδειξε και η Ρώμη 3. Έχουμε αυτή τη στιγμή 13 κανονισμούς, δύο οδηγίες για την δικαστική συνεργασία, ενώ εκκρεμούν πολλές προτάσεις, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Υπάρχουν κάποιες κατακαιρματισμένες αποσπασματικές διατάξεις διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που βρίσκονται σε πολλές οδηγίες ουσιαστικού δικαίου. Οπότε μπορούμε να καταλήξουμε γενικό στο συμπέρασμα ότι το ισχύον πλαίσιο έχει ε, έναν ευρύ αντίκτυπο και νομικό και πρακτικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια κενά εξαιτία του κατακαιρματισμού των κανόνων. Είναι κάπως ε, αποσπασματικό το πλαίσιο, ενώ μερικές φορές διαπιστώνουμε και επικάλυψη η επανάληψη των κανόνων. Τώρα, για να εντοπίσουμε τα κενά. Εντοπίσαμε τα κενά αυτού του κοινοτικού πλαισίου, καταρχήν αναλύοντα ε, τους επιμέρους κανονισμούς και το πεδίο εφαρμογή τους. Επίση, ε, διενεργήσαμε μια συστηματική ανάλυση του διεθνού ιδιωτικού δικαίου διαβάζοντας χειρίδια και βιβλιογραφία ε, είτε σε εθνικό είτε σε διεθνώς επίπεδο ε, για να βρούμε τις διάφορες διατάξεις και θεωρώ ότι ε, ο Ευρωπαίος Νομοθέτης θα πρέπει να επικεντρωθεί στα συστημικά κενά σε τομείς δηλαδή που είτε δεν υπάρχουν καθόλου κανόνες είτε υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες. Πού εντοπίζονται όμως αυτά τα κενά και πού χρειάζονται προσθήκες. Σε ό,τι αφορά ε, τομεί εκτό του οικογενειακού δικαίου, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν κανόνε για το, για το δίκαιο τη κυριότητα, για τα καταπιστεύματα, για τις οργα... Ε, σχέσεις των ε, οργανισμών, των, των εταιριών και σε θέματα οικονομικού δικαίου, θέματα διατησίας και άσκησης συλλογικών προσφυγών ελάχιστη καθόλου ρύθμιση δεν έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Τώρα, σε θέματα οικογενειακού δικαίου έχουμε ακόμη περισσότερα κένα. Κυρίω στο θέμα του γάμου, των καταχωρημένων σχέσεων ε, συμβίωση, ε, στα επώνυμα, υιοθεσία, συγγενική σχέση, ε, προστασία ενηλίκων ή καθεστώ και δικαιοπρακτική ικανότητα φυσικών προσώπων. Έχουμε κάποιου κανόνε για θέματα διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού με βάση το τη Ρώμη αλλά η Ρώμη δεν εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια, γιατί μόνο ε, λίγα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε αυτόν τον κανονισμό, γιατί εφαρμόστηκε η ενισχυμένη συνεργασία. Τώρα, βαίνουμε προς έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου γνήσιου ευρωπαϊκού κώδικα είναι ότι οι κανόνε αυτοί θα συμπεριληφθούν και θα συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο νομικό εργαλείο και μπορούμε με πολύ πιο συστηματικό τρόπο να τα προσεγγίζουμε, ξεκινώντας με τις γενικές αρχές και μετά προβλέποντας ε, συγκεκριμένα μέρη για τα επιμέρου ζητήματα. Θα πρέπει όμω να έχουμε υπόψη, και αυτό έδειξαν οι συζητήσεις ε, με τους συνομιλητές μας στα κράτη-μέλη ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν έχουμε όλοι την ίδια αντίληψη περί τι εστί κώδικας. Για παράδειγμα, στις συζητήσεις ε, με ε, ανθρώπους από τις χώρες του Common Law, ιδιαίτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι ακόμη και η ιδέα, η λέξη του κώδικα τους ε, απο, αποθαρρύνει, τους απομακρύνει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε κώδικα. Ίσως μερικοί είναι αρνητική ακόμη και στην αναφορά της λέξης κώδικα. Θα μπορούσαμε να πούμε απλώς πλαίσιο, αν ο όρος κώδικας ενοχλεί. Πολλές χώρες είναι υπέρ της διεύρυνσης του πλαισίου, αλλά δεν είναι όλες υπέρ αυτής της διεύρυνσης, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην προσέγγισή μας. Ούτε υπάρχει κάποια, κάποιος γενικός ορισμός για τους ε, υπερισχύοντες υποχρεωτικούς κανόνες ε, για διάφορες πολιτικές ή την εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου. Και εκεί υπάρχουν διστάμενες απόψεις και αντιλήψεις. Πρώτα λοιπόν θα πρέπει να ενοποιήσουμε την προσέγγιση μας και μετά να στραφούμε προς έναν πραγματικό ευρωπαϊκό κώδικα. Και υπάρχουν κενά και σε ζητήματα ουσιαστικού δικαίου. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ε, διαφορά σε ό,τι αφορά ζητήματα ουσιαστικού δικαίου, όπως είναι η παρέθετη μητρότητα, η συγγενική σχέση, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, οι καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης. Εκεί υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ουσιαστικού δικαίου των κρατών Δεν πρέπει να εμποδίζουμε τους κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, γιατί είδαμε κάτι που έχει να ε, αναγνωριστεί και θεσπιστεί σε μια χώρα θα πρέπει να έχει αποτελέσματα και σε άλλη χώρα. Αλλά για ορισμένου ευαίσθητου τομεί θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί ίσω δημιουργήσουμε κάποια προσκόμματα στην εφαρμογή των κανόνων διεθνού ιδιωτικού δικαίου. Τώρα, τι μέλη γενέστε, ποια είναι η ακολουθητέα πορεία. Μετά από συζητήσει που είχαμε και στην ομάδα εμπειρογνωμόνων μα, διαπιστώσαμε ότι ε, στο εγγύς μέλλον και μέσω πρόθεσμα θα πρέπει να γεμίσουμε κάποια κενά. Καταρχήν να δώσουμε έμφαση στο δίκαιο πλην του οικογενειακού. Ε, θέματα εταιρικού δικαίου, για παράδειγμα, η δικαίου της κυριότητας, ε, δεδομένης της κρίσης, θα ήταν προτεραιότητα τέτοια θέματα. Και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Επίσης, να δούμε την ομολογία του ΔΕΚ, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ακούσαμε τον Αντιπρόεδρο το πρωί θέματα επωνυμίας, ε, ε, συγγενικής σχέσης, ε, γάμων. Όλα αυτά είναι θέματα ιδιαίτερης προσοχής γιατί μερικές φορές πραγματικά δημιουργούν κολλήματα στην ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η αγαστή συνεργασία που χάνεται με την διάλεξη της Χάγης για την για το Διεθνέ Ιδιωτικό Δίκαιο. Γιατί, επαναλαμβάνω, ένα τμήμα των τομέων αυτών έχει καλυφθεί από τι διεθνεί συμβάσει και ο διάλογο με τη διάλεξη τη Χάγη για το Διεθνέ Ιδιωτικό Δίκαιο θα ήταν πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πώ θα γεμίσουμε αυτά τα κενά μέσω και μακροπρόθεσμα, μέσω μια σταδιακή ε, έγκριση ε, διαφόρων νομικών ή νομοθετικών διατάξεων. Και ίσως ε, όχι ταυτόχρονα όπως ε, έκαναν μερικές χώρες σε εθνικό επίπεδο. Τώρα και μακροπρόθεσμα είναι εφικτό ένα περιεκτικό πλαίσιο από τη στιγμή που θα πληρωθούν τα κενά σε ορισμένου τομεί και ενοποιηθούν κάποιοι ορισμοί και αναπτυχθούν κοινέ αντιλήψει για θέματα, θα είναι εφικτό να συνενώσουμε τους κανόνες και ίσως να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο εργαλείο και ενδεχομένως και σε έναν γνήσιο Ευρωπαϊκό Κώδικα Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Κράμερ. Πολύ ενδιαφέρουσα και η δική σας παρουσίαση. Και συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Νίκ Μπόζιτ, ελπίζω να το προφέρω σωστά, της ε, εταιρείας ICF ε, GHK από το Birmingham που θα μας παρουσιάσει τη μελέτη για το κόστος της μη ολοκλήρωσης της Ευρώπης και την προοπτική της ύπαρξης ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Παρακαλώ, κύριε Μπόζετ, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Λέγομαι Νίκ Μπόζιτ και είμαι εδώ γιατί Έχω εμπλακεί σε διάφορες μελέτες ε, αντικτύπου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάζοντας διάφορες προτάσεις. Ε, εδώ συμπεριλαμβάνουμε τα, τις περιουσιακές σχέσεις ε, συζύγων, κληρονομιές και διαθήκες. Αλλά αυτή η μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστιάζεται στο κόστος της μη ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε να δούμε τις διαστάσεις αυτού του κόστου, το κόστος στην κοινωνία, στα άτομα και στις επιχειρήσεις. Λόγω απουσίας ενός πραγματικά λειτουργικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ξέρω ότι εδώ περιστοιχίζουμε από νομοθέτες ε, στον τομέα της δικαιοσύνης και από νομομαθείς. Εγώ θα εξετάσω το πρόβλημα αυτό από διαφορετική σκοπιά από τη σκοπιά του οικονομολόγου και θα προσπαθήσω να το εδράσω σε κάποια παραδείγματα στο βαθμό του δυνατού. Σας έδωσα και ένα φυλάδιο στο οποίο σας παραπέμπω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βασιστεί σε, αυτά που είπε η προλαλήσασα, να δούμε τα κενά ποια είναι, να δούμε ποιες είναι οι διαστάσεις ε, του κόστους ε, της μη Ευρώπης, ειδικά στην ενιαία αγορά, για να δικαιολογήσουμε και να βρούμε την προστιθέμενη αξία μιας παρέμβασης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προσπαθήσουμε να δούμε σε ποιο βαθμό αυτό το κόστος μπορεί να εξοικονομηθεί, να μην ταπανηθεί, δηλαδή μέσω της χρήσης του ιδιωτικού δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου. Λοιπόν, αυτή είναι μια μελέτη, θα σας την παρουσιάσω και θα ακούσω και τις παρατηρήσεις σας, τις οποίες θα λάβω υπόψη. Λοιπόν, το κόστος πιο... της μη Ευρώπης είναι προκύπτει από το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικά νομικά καθεστώτα ε, στι ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιδιωτικό διεθνέ δίκαιο, όπως ακούσαμε, ορίζεται, δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτόν τον ορισμό, μπορούμε να το περιορίσουμε σε θέματα του ποιος ε, εκδικάζει, στην αναγνώριση των αποφάσεων, αλλά μπορεί να περιέχει και υπιότερα μέτρα, ούτω ώστε να μειωθεί αυτό το κόστος τη μη Ευρώπης. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα ωφέλη της κωδικοποίησης ενός μελλοντικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Για να σκεφτούμε λοιπόν καταρχάς ποιο είναι το κόστος και πώς μπορεί να μετριαστεί. Υπάρχει κόστος για τους πολίτες, ακόμη και για τους ανήλικου από την παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας του και λόγω αβεβαιοτήτων στις νομικές σχέσεις, ε, καθυστερήσεων και πιθανού, πιθανής παραβίασης των δικαιωμάτων σε οικογενειακά θέματα. Υπάρχει κόστος λόγω μεγαλύτερων καθυστερήσεων, αβεβαιότητας ε, και ψυχολογικής, ε, ψυχολογικών προβλημάτων για τους πολίτες. Επίσης, ε, υψηλότερο κόστο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες λόγω διαφορών στα νομικά καθεστώτα. Επίσης, ε, ε, επηρεάζουν αυτό τις διασυνορικές συναλλαγέ επιχειρήσεων με καταναλωτέ. Και αυτό αυξάνει το κόστος. Επίσης, αυξάνεται το κόστος παραγωγής και επένδυσης λόγω διαφορών των νομικών καθεστώτων. Αυτό επηρεάζει τον τόπο εγκατάστασης και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων όταν είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικό κράτος μέλος. Αυτές οι διαφορές μπορεί να συνεισφέρουν και να δημιουργούσουν τριβές, να αποθαρρύνουν τον κόσμο, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και έτσι να αυξηθεί το κόστος ε, παραγωγής ε, αγαθών και, και υπηρεσιών λόγω διαφορών στα κράτη-μέλη. Ε, έτσι Και γιατί θα έχουμε χαμηλότερη κινητικότητα το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι ένα επιπλέον κόστος για, την, για το σχεδιασμό της ε, συναλλαγής ή της ενοχής. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και ένα διεθνές ε, ζευγάρι που μπορεί να ετοιμάζεται να παντρευτεί ή μια εταιρεία που ετοιμάζεται να κάνει μια επένδυση σε έναν άλλο Επίση, Επίσης το επιπλέον κόστος και η καθυστέρηση στις νομικές ε, διαδικασίες συμπεριλαμβάνει και το κόστος για την πληρωμή των ε, νομικών ε, που θα ασχοληθούν με αυτές τις διαφορές λόγω των διαφορετικών καθεστώτων στα κρατη Είναι ε, ακριβό το να συγκεράσουμε τις διαφορές, το ξέρουμε. Και μερικές φορές και τα άτομα και οι επιχειρήσεις προτιμούν να υποφέρουν από το να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ε, δεν κάνουν, δεν ασκούν λοιπόν αγωγές. Υπάρχει το κόστος της νομικής αβεβαιότητας, το ψυχολογικό κόστος και κυρίως πιθανές επιπτώσεις στο πιο αδύναμο μέρος. Ε, υπάρχει και το κόστος του διαφυγόντος κέρδους. Ε, γιατί κάποιος δεν θα προβεί σε μια συναλλαγή, σε μια ενοχή, σε μια σύμβαση και ένας καταναλωτής μπορεί να επιλέξει να πληρώσει περισσότερο για το ίδιο πράγμα, ίδιες συνθήκες κτλ. αντί να προσφύγει ε, σε κάποιο αγαθό ή κάποια υπηρεσία από ένα κρατός μέλος. Μερικές φορές πρόκειται για τον ίδιο ε, πάροχο, ή για τον ίδιο προμηθευτή. Επιλέγουμε όμως ε, με βάση το κράτος μέλος και όχι με βάση την τιμή. Ακόμα και όταν λαμβάνουμε τις διαφορές ε, του ΦΠΑ για το ίδιο προϊόν και για τον ίδιο προμηθευτή. Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει αυτές τις διαφορές και αυτό προσθέτει δισεκατομμύρια στο κόστος της μη Ευρώπης εντός αγωγικών. Ποιο είναι το κόστος για τους πολίτες σε οικογενειακά θέματα και υποθέσεις. Όλο και περισσότερα διεθνή ζευγάρια έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ μεταξύ αυτών είμαι. Ε, γιατί η γυναίκα μου είναι Γαλλίδα. Υπάρχουν ε, επιπλέον ε, νομικές δαπάνες, ψυχολογικό κόστος, γιατί είναι πιο ακριβό το να λυθούν διαφορές σε ορισμένες οικογένειες ε, που συνδέονται με το γάμο, τις ε, γονικές ευθύνες, το διαζύγιο, τις ε, κληρονομιές και τις διαθήκες. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το υψηλότερο κόστος για, τις, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις είναι απρόθυμες να συναλλαχθούν διασυνοριακά λόγω του κόστους προσαρμογής στη διασυνορική δραστηριότητα και λόγω των εθνικών ε, νόμων προστασίας των καταναλωτών που επισύρει αβεβαιότητα σε περίπτωση διαφορών. Ε, παράλληλα και οι καταναλωτές είναι απρόθυμοι να προβούν σε τέτοιες συναλλαγές για τους ίδιους λόγους, αβεβαιότητα για το αν θα υπάρξει δυνατότητα ένδικων, άσκησης ένδικων μέσων. Αυτό οδηγεί σε διαφορετικέ τιμέ για τα ίδια αγαθά και τι ίδιε υπηρεσίες, όπως εξήγησα, ακόμα και όταν προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή υπάροχο. Τώρα, στον τομέα τη αφαιρεγκαιότητα. οι επιχειρήσει μπορεί να είναι απρόθυμες να εγκατασταθούν στο εξωτερικό λόγω αβεβαιοτήτων για τι διαδικασίε αφαιρεγκαιότητα. Και οι πιθανοί πιστωτέ μπορεί να μην θέλουν να προχωρήσουν σε συναλλαγές με ξένε επιχειρήσει, γιατί μπορεί να θεωρήσουν ότι αυτοί θα υποβιβαστούν σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας και δεν θα πληρωθούν πρώτοι. Σε περίπτωση είτε αφαιρεγγιότητας είτε πτώχευσης κτλ. Επομένως, όλες αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες ε, δεν γίνονται με το βέλτιστο τρόπο. Και αυτό επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις τρίτες ε, χώρες. Ακόμα και στην αγορά των δημοσίων προμηθειών έχουμε τα ίδια προβλήματα. Αυτό έχει συνέπειες. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία. Και επιπλέον οδηγούν σε ανισορροπίες στην αγορά εργασίας. Έχουμε προβλήματα σε ορισμένα κρατημέλη, σε ορισμένου τομεί, ε, σε ό,τι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση εργατικών χεριών. Υπάρχει λοιπόν πολύ ψηλό κόστος εδώ. Εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά που είπε και η προλαλήσασα. Δεν θέλω να διατρέξω αυτούς τους τομείς, θέλω να αγγίξω ε, λίγο το παράδειγμα των περιουσιακών σχέσεων συζύγων. Υπάρχουν διαφορές στα νομικά καθεστώτα των κρατών μελών. Το βασικό πρόβλημα είναι η ατελής και αναποτελεσματική, ο ατελής και αναποτελεσματικός χειρισμός της εκαθάρισης των διεθνών περιουσιακών καθεστώτων. Αν η οικογένεια έχει ας πούμε, περιουσιακά στοιχεία σε διαφορετικά κράτη-μέλη, αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι χρειάζεται. Ποιο επηρεάζεται. Κυρίω ο πρώην σύζυγος ή χείρος, η σύντροφος ε, του διεθνού ζευγαριού σε περίπτωση ε, διαζυγίου ή θανάτου ποιες είναι οι επιπτώσεις, είναι ψυχολογικό άκθος, ε, κόστος ε, και καθυστερήσεις. Προσπαθούμε, να προσμετρήσουμε όλο, όλο αυτό το κόστος. Ποια είναι η κλίμακα του προβλήματος. Υπάρχουν 122 εκατομμύρια γάμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ καλύπτουμε και τις επίσημες σχέσεις και 20 εκατομμύρια έχουν και ένα διεθνέ στοιχείο. Δηλαδή ε, σύντροφοι από διαφορετικά κρατημέλη ή ο ένας από τους δύο συντρόφους είναι από τρίτη χώρα. Πολλά ζευγάρια παρά τα προβλήματα με τη μετακίνηση ε, μπορεί να ζουν σε άλλη χώρα από τη δική τους. Μπορεί να μην ξέρουν ε, τι να αντιμετωπίσουν σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους. Πολλοί έχουν ε, και περιουσία στο εξωτερικό. Μπορεί να αυξήσει αυτό τις δυσκολίες. Και δυστυχώς, ή μάλλον ευτυχώς, υπάρχουν γάμοι. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και διαζύγια. Και βεβαίως υπάρχουν και χωρισμοί λόγω θανάτου. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία που σας δίνω είναι αρκετά αξιόπιστα. Το πρόβλημα είναι όταν μπούμε σε, στις λεπτομέρειες, όταν προσπαθούμε να δούμε ποιο είναι το κόστος σε κάθε περίπτωση. Ποιο είναι το είδος του κόστους. Όταν κανείς παντρεύεται ή έχει μια επίσημη σχέση, είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσει τα δικαιώματά του. Μερικές φορές θα υπάρξει νομικό κόστος μέσα στο γάμο όταν τα δικαιώματα των συζύγων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να περιορίζονται. Μπορεί να υπάρχει επιπλέον κόστος σε περίπτωση διαζυγίου. Ειδικά όταν δεν είναι συνετικό το διαζύγιο. Και επιπλέον, επιπλέον κόστος κατά το θάνατο ενό συζύγου όταν χρειάζονται διευκρινήσει για τα δικαιώματα, ειδικά σε ό,τι αφορά την περιουσία και ειδικά όταν υπάρχουν διαφορές για την περιουσία. Σας έχω ετοιμάσει και ένα πίνακα που δείχνει την προσέγγισή μας ε, και στο πώ στο πώς μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε ε, το κόστος αυτό. Οι νομομαθεί μου λένε πόσο συχνά ε, προκύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα και τι κοστίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα στη συγκεκριμένη φάση, όταν έχουμε διεθνείς γάμους, και τα άτομα αυτά ζουν στο εξωτερικό ή έχουν περισσιακά στοιχεία στο εσωτερικό, κάνουμε μια εκτίμηση. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι το κόστος. Κάνουμε κάποιες υποθέσεις βέβαια εδώ. Αλλά προσπαθούμε να έχουμε, κάνουμε συντηρητικές υποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, Βάζουμε μόνο το, το άμεσο κόστος εδώ. Ε, δεν βάζουμε το έμεσο κόστος. Αν το βάζαμε θα ήταν πολύ ψηλότερο το κόστος. Στη μελέτη αντικτύπου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβαμε υπόψη τις προτάσεις και εκτιμήσαμε το κόστος τιμή Ευρώπης και πώς μπορεί να μειωθεί με τις προτάσεις που είναι τώρα επιτάπητος. Τώρα, η δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια αντίστοιχη προσέγγιση στους άλλους τομείς που ανεφέρθηκαν και στα άλλα κενά που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπόζετ γιατί μας ε, σκιαγραφίσετε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πλήρη επίγνωση το ότι υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα και ένας τεράστιος χώρος όπου υπάρχει δυνατότητα ε, ενοποίησης, εναρμόνισης ε, κοινών διατάξεων και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα μειωθεί και το οικονομικό αλλά κυρίως το συναισθηματικό κόστος γιατί υπάρχουν δυνατότητες διευκόλυνσης ε, της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των διαφόρων συναλλαγών των πολιτών των διαφόρων καταστάσεων. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα βέβαια η γνώμη και των εθνικών βουλευτών για τα θέματα αυτά. Έχουμε τώρα προβλέψει ένα, χρόνο, ένα χρόνο για συζήτηση, για ερωταπαντήσεις. Δεν έχω λάβει επίσημα κανένα αίτημα για το λόγο. κύριος Μασίπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι Ευρωβουλευτής και μέλος Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Για μένα λοιπόν ήταν πολύ σημαντική αυτή η ευκαιρία και άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρωινό τμήμα της και το απόγευμα θα προτιμήσω να μην παραστώ σε άρισμα υποχρεώσεις και να ακούσω τον πρώην Ευρωβουλευτή Κουρτ Λέχνερ και την κυρία Αλεξάνδρε Τάιν. Από όσα άκουσα σήμερα Κάτι που μου τράβηξε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι κάτι που επιδιώκουμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η προσπάθεια να μειώσουμε το κόστος εξαιτίας της ε, έλλειψης της ελευθερίας, της ταχύτητας ε, και της ευκολίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συμβολογράφος ο κύριος Πρέγερ μας είπε, γιατί και εγώ ήμουν για πολλά χρόνια δικηγόρος, μέχρι το 2004 εξελάγει Ευρωβουλευτής, και έχω και εγώ πολύ αρνητική πείρα από το ίδιο μου το επάγγελμα. Όταν ήμουν στη δεκαετία του 60 νέος δικηγόρος, μιλάμε για μισό αιώνα πριν δηλαδή και πρώτη φορά ε, μετά την, την, που κληρονόμησε το γραφείο του πατέρα μου και άρχισα να εργάζομαι, διαπίστωσα ότι τα περισσότερα δικηγορικά γραφεία στην ε, πόλη που ασκούσα εγώ το επάγγελμα ήταν ε, ορκισμένοι εχθροί της διαμεσολάβησης. Προτιμούσαν τις δίκες. Ε, τότε δεν ήταν και πολλές οι δίκες, αλλά αυτό επιδίωκαν οι δικηγόροι. Ήταν υπέρ της ε, ένδικης αντιπαράθεσης. Πέρασε τώρα μισός αιώνας και παρακολούθησα όλο το πανόραμα της δικηγορίας και της πολιτικής και διαπίστωσα ότι υπήρξε κάποια εξέλιξη. Γιατί εξαιτίας της περιπλοκότητας του δικαίου και του πληθωρισμού του δικαίου και των δικών άλλαξε κάπως το τοπίο και άλλαξε κάπως η νοοτροπία διαπιστώνουμε ότι πολύ περισσότερο το σημαντικότερο είναι η συνδιαλλαγή, ε, είτε δικαστικός συμβιβασμός, είτε ο εξωδικαστικός μέσω διαμεσολάβησης. Ο κύριος Πρέγερ λοιπόν ρώτησε το κρατήριο «Πιστεύετε ότι χάρη στη διαμεσολάβηση θα μειωθεί το κόστος το δικηγορικό» από τη στιγμή που θεσπίστηκε στην Ευρώπη. Το αμερικανικό σύστημα δικηγορικών αμοιβών και εξόδων και μπορούν οι δικηγόροι να χρεώνουν ε, την ώρα της απασχόλησής τους και μερικές φορές και το λεπτό και το δευτερόλεπτο, διαπιστώνουμε ότι σίγουρα ε, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά των αμοιβών, ε, είτε έχουμε δίκη είτε διαμεσολάβηση από τη στιγμή που συμμετέχουν δικηγόροι. Πάντως θα πρέπει και οι Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να πιάσουν τον τάβρο από τα κέρατα, όπως λέμε στην Ισπανία, και να υιοθετήσουν ένα σύστημα που θα είναι πραγματικά ελκυστικό. Και να είναι ελκυστική διαμεσολάβηση όχι μόνο εκ του αποτελέσματος, όχι μόνο γιατί ε, είναι αναγκαιότητα η διδατολογική προετοιμασία και η ηθική προετοιμασία των διαμεσολαβητών, αλλά γιατί τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν και ρυθμίσεις και φορολογικές διατάξεις που να εξωθεί, να παροτρύνει και τους ίδιους δικηγόρους να στρέφονται προς τη διαμεσολάβηση και να την αναζητούν ως ε, πρώτη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων και των διαφορών. Ακούσαμε και μία καθηγήτρια από τον Μπίρμιχαμ. Και εγώ είχα μια δύσκολη περίπτωση διαμεσολάβηση και εγω ειχα μια δυσκολη περιπτωση διαμεσολαβηση και συνδιαλογη με τον Μπίρμιχαμ. Και μάλιστα καταφέραμε την συμφιλίωση σε μια τρίτη χώρα τελικά, γιατί ήταν πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο δαπανηρή η δικηγορική αμοιβή των δικηγόρων στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Πράγερ πραγματικά άγγιξε το ευαίσθητο σημείο για το πώς μπορούμε να ανάξουμε την πραγματικότητα και την οτροπία υπέρ της διαμεσολάβησης. και θα πρέπει μαζί με τους δικηγόρους και τις χώρες μέλη να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε μια πολύ πιο εύκολη επικοινωνιακή Ευρώπη όπου οι διασυνοριακές σχέσεις θα είναι πολύ πιο εύκολες, θα πρέπει να λύσουμε πρώτα αυτό το κέριο ζήτημα. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε σήμερα εδώ και μας εθαρρύνατε. Γιατί αυτά που θα πείτε και που θα σημειωθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης θα δώσουν κίνητρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επιβάλλουμε κάποια κριτήρια ε, ταχύτητας ε, και ευληγησίες που είναι χρήσιμα όχι μόνο για το επάγγελμα του δικηγόρου, αλλά πολύ πιο χρήσιμα θα είναι για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μασίπ για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Μασίπ είναι Ισπανός Ευρωβουλευτής όπως ακούσαμε. Δεν ξέρω αν έχετε υπόλοιποι ερωτήσεις, παρατηρήσεις, ε, σχόλια για το μέχρι τώρα μέρος της συζήτησης. Δεν βλέπω να θέλει κανείς το λόγο, οπότε μπορούμε να περάσουμε σε λίγο στις επόμενες μας παρεμβάσεις. Θα ήθελα να σας ε, επισημάνω ότι μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μας ε, τα έγγραφα του σημερινού σεμιναρίου. Περνάμε τώρα στις ακόλουθες ομιλίες. Θέμα του σημείου αυτού θα είναι ο κανονισμός 2 και οι οδηγίες για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Έχουμε δύο καλεσμένους, δύο εμπειρογνώμονες. Πρώτα από το Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελτ. Ο καθηγητής Άδικας Στάουτιγκερ. Κύριε Στάλφη, ε, τα ε, οδικά ατυχήματα με διεθνή διάσταση στην εσωτερική αγορά είναι όλο και συχνότερα και στόχος του Ευρωπαίου νομοθέτη θα, ή πρέπει να είναι η νομική ενιαιότητα, ασφάλεια και μια ισορροπία μεταξύ των αντικρουωμένων συμφερόντων. Έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κατά την εμπειρία μου μόνο μερικά. Να αναφέρω μία απλή περίπτωση. Κάποιος λοιπόν, ο οποίος έχει το κέντρο συμφερόντου στο, στη Γερμανία, εάν λοιπόν αυτό το άτομο πάει στο Βέλγιο και αν εδώ στο Βέλγιο ε, πάθει ένα ατύχημα, οδικό ατύχημα, τίθεται το ερώτημα σε, σε ποια χώρα θα προσφύγει κατά ποιου. Όταν θα γυρίσει στη Γερμανία θα μπορούσε να σκεφτεί να προσφύγει κατά του Βέλγου οδηγού και της ασφάλειάς του. Αλλά αυτό δεν έχει έννοια. Ε, έννοια έχει κυρίως ε, να μην στραφεί κατά του ε, ε, διαπράξαντος το δίχημα, αλλά κατά της ασφάλισης του. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτός ο, ο ενάγων, ο οποίος ζει στην ε, Γερμανία, μπορεί να προσφύγει όχι μόνο στο Βέλγιο κατά της υποχρεωτικής ασφάλισης ε, του Βέλγου, αλλά και στη Γερμανία. Αυτό λέει η Σύμβαση Βρυξέλλες 1. Και η μεταρρύθμισή της, ο νέος κανονισμός επιτρέπει στους ενάγοντες να προσφύγουν στην χώρα από την οποία προέρχονται κατά ε, του ε, διαπράξαντος το ατύχημα μέσω της ασφάλισής του στην ε, Γερμανία. Αυτό συνέβη και ε, σε σχέση με την Δανία και ισχύει, ισχύει και με την σύμβαση του Λουγκάνο. Πώς έχει όμως το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Όταν θα γίνει η προσφυγή στην Γερμανία τότε το γερμανικό δικαστήριο θα εφαρμόσει τον κανονισμό Ρώμη 2. Όμως δεν ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή η σύμβαση. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν την οδική σύμβαση της Χάγης. Η Δανία εφαρμόζει την δική της διεθνή σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Έχουμε λοιπόν ε, ένα αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες για αυτέ τι περιπτώσεις. Αλλά δυστυχώ οι τρει δεν πηγαίνουν προ την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ω εξή. Υπάρχουν τρει πηγέ δικαίου για το ιδιωτικό διεθνέ που μπορεί να καταλήξουν σε διαφορετικές αποφάσεις επί της ουσίας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει κανείς forum shopping, επιλογή δικαιοδοσίας. Δηλαδή, μπορεί να προσφύγει κατά της ασφάλειας όχι μόνο στη χώρα προέλευσής του αλλά και στη χώρα όπου έχει την βάση του η ασφαλιστική εταιρεία. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιήσει την ε, σύμβαση της Χάγης, τη σύμβαση των, της Ρώμης ή την ε, Δανέζικη σύμβαση όπως σας είπα. Είπαμε λοιπόν ότι στόχος μας πρέπει να είναι η ενιαία αντιμετώπιση. Δεν έχει επιτευχθεί λοιπόν σε περίπτωση ιδιωτικού δικαίου. Τι σημαίνει αυτό για την ε, νομική ασφάλεια. Εάν γίνει η δίκη στην ε, Γερμανία, τότε ο Ενάγων κάνει απευθεία ε, προσφυγή κατά του Βέλγου ασφαλιστή, κατά των βελγικών ασφαλιών. Αλλά σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε τα εξή. Το γερμανικό δικαστήριο είναι διεθνώ αρμόδιο, αλλά πρέπει μέσω της Ρώμης 2 να εφαρμόσει δίκαιο άλλης χώρας. Τι σημαίνει δίκαιο άλλης χώρας ε, σε μια τέτοια περίπτωση. Είναι πολύ διαφορετική η ερμηνεία ε, του ξένου δικαίου. Ε, στη Γερμανία θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά το ε, ξένο δίκαιο. Αλλά αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες. Υπάρχει διαφορετική ε, δικονομική συμπεριφορά. Όταν λοιπόν ε, παίζει ρόλο το ξένο δίκαιο είναι πολύ πιο ε, ακριβή η διαδικασία και κρατάει πολύ περισσότερο. Επιπλέον ένα γερμανικό δικαστήριο όταν εφαρμόζει το ξένο δίκαιο σε τελευταία ανάλυση είναι υποχρεωμένο να δώσει την αρμοδιότητά του να αποδώσει την αρμοδιότητά του σε έναν εμπειρογνώμονα. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα λάθους όταν εφαρμόζεται ένα ξένο δίκαιο από ένα δικαστήριο που δεν είναι συνηθισμένο να εφαρμόζει ξένο δίκαιο. Και ποια είναι η προβλεψιμότητα για το τι απόφαση θα υπάρξει. Ούτε για τους ε, δικηγόρους στην Γερμανία δεν είναι μεγάλη, ούτε για τους εμπλεκομένους. Ξέρετε ότι με βάση την Ρώμη 2, ένα γερμανικό δικαστήριο, με βάση το αιτιολογικό 33, μπορεί το γερμανικό δικαστήριο να τροποποιήσει την εφαρμογή εξωτερικού δικαίου και υπάρχουν και επιφυλάξεις ε, δημόσιας τάξης. Άρα η ε, έκβαση μιας διαδικασίας ενός γερμανικού δικαστηρίου που εφαρμόζει ξένο δίκαιο δεν είναι προβλέψιμη. Αυτό σημαίνει δεν είναι δεδομένη ούτε καν η νομική ασφάλεια. Αυτό οδηγεί στην εξή συνολική εικόνα. Βεβαίως ο ενάγων μπορεί να προσφύγει κατά του ξένου, ε, της ξένης ασφάλειας, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί ξένο δίκαιο και αυτό οδηγεί σε ακριβότερη διαδικασία, πιο μακροσκελή διαδικασία, γιατί πρέπει να ερμηνευτεί το ξένο δίκαιο και δεν υπάρχει προβλεψιμότητα για το αποτέλεσμα. Τι δυνατότητα θα είχαμε να εξεύρουμε άλλη λύση. Στο έγγραφό μου προτείνω το εξή. Φυσικά, έχουμε δυνατότητα ε, να επιλέξει, έχει δυνατότητα να επιλέξει ο ενάγων που να απευθυνθεί. Μπορεί να προσφύγει στη χώρα του κατά της ξένης ασφάλειας. Αυτό ε, συνδυάζεται, συνάδει με το δικαίωμα καταναλωτή. Ένας καταναλωτής μπορεί να έχει το δικαίωμα να ε, χρησιμοποιήσει τη διαδικασία που θεωρεί ότι είναι πιο επωφελής για αυτόν. Αλλά Εάν ένα γερμανικό δικαστήριο είναι διεθνώς αρμόδιο, είναι προφανές ότι για την απευθείας απέτηση έναντι ενός ξένου ε, εναγωμένου είναι χρήσιμο να μπορεί να εφαρμόζεται το εσωτερικό δίκαιο, το lex fori, διότι ένα γερμανικό δικαστήριο πρέπει να βασίζεται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα έπρεπε να μπορεί οποιοδήποτε δικαστήριο να προσφύγει κατά ενός ε, εξωτερικού εναγωμένου. Αυτό μπορεί να γίνει γιατί και στην Ρώμη 2 και στην Σύμβαση της Χάγης υπάρχει μια ειδική διάταξη που το επιτρέπει αυτό σε τελευταία ανάλυση. Θα ήταν λοιπόν μόνο μια συμπλήρωση, μια εφαρμογή της νομολογίας όπως έχει μέχρι τώρα. Και τι επιπτώσεις θα είχαμε. Εάν τώρα ένα εσωτερικό δικαστήριο όταν εναχθεί, όταν υπάρξει εναγωγή, ε, ε, όταν υπάρξει προσφυγή σε αυτό, εφαρμόσει το εσωτερικό δίκαιο. Πρώτον λοιπόν δεν χρειάζεται εμπειρογνώμων, είναι φθηνότερη δίκη, ταχύτερη και ε, είναι μικρότερη η πιθανότητα λάθους. Το αποτέλεσμα λοιπόν θα ήταν επίσης πιο προβλέψιμο για όλους τους εμπλεκομένους, για τους δικηγόρους. Οπότε θα υπήρχε και ενιαιότητα δικαίου και νομική ασφάλεια. Και, όπως ξέρετε, επίσης, ο ενάγων ζει σε μια συγκεκριμένη χώρα και είναι πολύ λογικό να εφαρμόζεται η αρχή της χώρας. Είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει αποζημίωση με βάση το δίκαιο του περιβάλλοντος όπου ζει το θύμα θα μπορούσε κανείς να αντιπεί ότι για τις επιχειρήσεις δεν είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο, διότι θα έπρεπε ενδεχομένως να πληρώσουν περισσότερο. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Ο κανονισμός, ο διακανονισμός ενός τέτοιου ατυχήματος, με βάση το δίκαιο της χώρας όπου ζει ο ενάγων, δεν είναι κατά ανάγκη ακριβότερος από τις άλλες εναλλακτικές λύσεις. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση υπάρχει ε, το κόστος της ε, ε, ερμηνείας του δικαίου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ακριβότερη η επίλυση της διαφοράς. Γι' αυτό θα ήταν δυνατόν να αναλάβουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες, να προτιμήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες μια τέτοια λύση, γιατί είναι προβλέψιμο το κόστος της, μπορεί να υπολογιστεί και άρα μπορεί να κάνουν αντασφάλιση. Άρα έχουν μια καθαρά μαθηματική ε, λύση σε ένα πρόβλημα για το πώς θα διασφαλίσουν την επιχείρησή τους, άρα οικονομικά είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Τι πρέπει να κάνουμε πολιτικά. Είναι δύσκολο να επιβάλλουμε σε όλα τα κράτη να ακολουθήσουν την Ρώμη 2 και τα κράτη που προτιμούν ε, το μοντέλο της Χάγης δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθούν να σταματήσουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για τις απευθείας απαιτήσει να υπάρξει μια ειδική ρύθμιση μέσω ενός κανονισμού με βάση τον οποίο όταν ο ενάγων προσφεύγει στην χώρα καταγωγής του κατά της υποχρεωτικής ασφάλισης που είναι σε άλλη χώρα, τότε να εφαρμόζεται η αρχή του lex fori, δηλαδή να εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας όπου διαμένει ο ενάγων. Θα ήταν λοιπόν μια ειδική ρύθμιση για αυτές τις ειδικές περιπτώσεις μόνο για την περίπτωση όπου το κέντρο ενδιαφερόντων, η χώρα διαμονής, είναι σε ένα κράτος μέλος και η ασφάλεια σε ένα άλλο κράτος μέλος. Είναι θέμα λοιπόν ενιαίας αγοράς και ελπίζω οι Ευρωπαίοι νομοθέτες να έχουν την αποφασιστικότητα να επιλύσουν το θέμα αυτό, γιατί σε τελευταία ανάλυση αυτό θα αφορούσε μόνο ένα μικρό τμήμα των περιπτώσεων και θα είχαμε λοιπόν ενιαιότητα του δικαίου, νομική ασφάλεια και ε, λογική προβλεψιμότητα για όλους τους εμπλεκομένους, δηλαδή θα εποφελούνταν και οι ενάγοντες αλλά και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη δεύτερη μας ομιλήτρια για το θέμα αυτό, την κυρία Τζένι Παπέτας από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιχαμ. Uh, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που με προσκάλεσε για να μιλήσω σήμερα εδώ. Παρόμοιο είναι το θέμα μου με του καθηγητή Στόντιγκερ. Φυσικά το θέμα είναι τα διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα και το δίκαιο που εφαρμόζεται για να επιληθούν οι διαφορές ε, σε αυτά τα ατυχήματα. Θα ήθελα να για τη σχέση ε, μεταξύ του Ρώμη 2, τη Σύμβαση της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο για τα τροχαία ατυχήματα και την οδηγία για τα, τις ασφαλιστικές εταιρείε. Έχω δέκα λεφτά στη διάθεσή μου και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις της συνύπαρξης και της ταυτόχρονης λειτουργίας αυτών των τριών καθεστώτων. Επομένως, θα αποπειραθώ απλώς να σας μιλήσω για τη σχέση μεταξύ των τριών αυτών καθεστώτων και θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα για την περιπλοκότητα και την αβεβαιότητα που προκύπτει εν μέρη από τους κανόνες του ίδιους και εν μέρη από την αλληλεπίδραση των καθεστώτων. Θα καταλήξω λέγοντας ε, κατά τη γνώμη μου τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Παράδοξο είναι ότι ο κύριος Στόντιγκερ ε, έχουμε φτάσει στο ίδιο συμπέρασμα, παρότι φτάσαμε στο ίδιο συμπέρασμα μέσω διαφορετικών οδών. Τα τροχαία ατυχήματα είναι των αρχιετυπικών μη ενοχικών υποχρεώσεων και συχνά φορούν α, απλές υποθέσεις, απλά γεγονότα. Όμως σε μια διασυνοριακή υπόθεση μπορεί να αυξηθεί η περιπλοκότητα των υποθέσεων αυτών για να δούμε ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Φανταστείτε το εξή σενάριο. Μία Γαλλίδα που μένει μόνιμα στο Παρίσι θέλει να ταξιδέψει για δουλειές στο Τρίερ και πάει δηλαδή στα σύνορα με τη Γερμανία κοντά στο Λουξεμβούργο. Ε, πετάει στο Λουξεμβούργο Οι συνάδελφοί της έχουν κλείσει το ταξίδι. Στο ταξίδι της, ε, ενώ είχε πάρει ταξί για τη Γερμανία, ο ταξιτζής ε, προσκούησε ένα δέντρο και η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά. Ασκεί ε, αγωγή εναντίον του, της ασφαλιστικής εταιρείας του ταξιτζή σε γαλλικό δικαστήριο ο, φυσικά ο ταξιζής είναι Λουξεμβούργιος, βρίσκεται στο Λουξεμβούργιο και το ερώτημα για το γαλλικό δικαστήριο είναι ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο με το οποίο θα εκδικαστεί η υπόθεση. Ένα καλό σήμα είναι το Ρώμη 2. Το άρθρο 1 της Ρώμης 2 λέει ότι το Ρώμη 2 ε, ισχύει μόνο σε μη συμβατικές υποχρεώσεις. Αυτό το μη συμβατικές πρέπει να έχει αυτόνομη έννοια και θα πρέπει να εφαρμόζεται και να ερμηνεύεται τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν υπάρχει αμφιβολία για την απέτηση, τότε μπορούμε, ας πούμε, να υποθέσουμε ότι το Ρώμη 2 ισχύει για, τον, για την υπόθεση αυτή. Το άρθρο 28 του Ρώμη 2 λέει ε, ότι η Γαλλία, αφού έχει προσυπογράψει τη Χάγη και τη στιγμή της υιοθέτηση υιοθέτησης ε, της, του Ρώμη 2, η εφαρμογή της σύμβασης ε, δεν θα πρέπει όμως να εμποδιστεί από, την, από τον κανονισμό και μπορεί να εφαρμόσει το, τη σύμβαση. Ε, στο άρθρο 1 η σύμβαση λέει ότι ε, έτσι επιλύονται αυτές οι διαφορές. Αυτό όμως δεν έχει αυτόνομη σημασία. Σε κάθε φάση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς κανόνες ε, ταξινόμησης της αγωγής. Ο ορισμός του non-contractual, του μη συμβατικό, επηρεάζεται από τους ορισμούς που χρησιμοποιεί το 2. Αν το Γαλλικό Δικαστήριο θεωρεί ότι η φύση της αγωγής είναι α, συμβατική και όχι μη συμβατική, με βάση τους εσωτερικούς κανόνες πριν της Ρώμης, τότε δεν ισχύει η Σύμβαση της Χάγης για την αγωγή αυτή. Αν ο ορισμός ε, ισχύει με βάση το Ρώμη 2, τότε ισχύει, ή μάλλον όχι, μπορεί να ισχύει ε, η Σύμβαση της Χάγης και άρα υπάρχει αμφισβηβολία εδώ. Λοιπόν, άρθρο 1, ορισμός ε, και πώς επηρεάζεται από το Ρώμη 2 για τις ε, συμβατικές υποχρεώσεις. Στο άρθρο 4F της Σύμβασης, το εφαρμοστέο ε, δίκαιο είναι το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Γιατί είναι, ε, εκεί έχει καταχωρηθεί το όχημα, το οποίο έχει εμπλακεί στο ατύχημα και, το, και ο επιβάτης που είναι θύμα διαμένει εκτός του κράτους αυτού όπου γίνεται το ατύχημα το εφαρμοστέο δίκαιο ε, είναι το ίδιο με την κατοικία του, του ενάγοντα. Αν ε, το γερμανικό δίκαιο είναι αυτό που ρυθμίζει την αποζημίωση, τότε ε, αν λάβουμε υπόψη μας και το δίκαιο του Λουξεμβούργου μπορεί να δημιουργηθεί α, forum shopping. Και με βάση το Ρώμη 2 θα ισχύσει το γερμανικό δίκαιο. Αν θεωρήσουμε ότι το Γαλλικό Δικαστήριο που εφαρμόζει τη Σύμβαση τη Χάγη τότε θεωρεί ότι το Λουξεμβούργιο δίκαιο ισχύει, το επόμενο ερώτημα είναι πώ μπορεί να επηρεαστεί από την οδηγία για τι ασφάλειε αυτοκινήτων. Το άρθρο 14 τη οδηγία αυτής είναι σημαντικό, το οποίο λέει ότι ο ασφαλιστή θα πρέπει να καλύψει τα, τα έξοδα με, και θα πρέπει να, καλύψει, να τα καλύψει με γενναιόδωρο τρόπο. Αυτό ισχύει παρά το Ρώμη 2 και τη σύμβαση του Χάγη. Το Ρώμη 2 θεωρεί ότι μπορεί να επιλεγεί δικαστήριο στο άρθρο 16 και προβλέπει ότι οι κανόνες για την επιλογή του δικαστηρίου ε, ε, ρυθμίζονται με άρθρο το 27. Ε, η οδηγία για την ασφάλεια των αυτοκινήτων ε, έχει πρωτοκαθεδρία σε σχέση με το Ρώμη 2. Σε σχέση με τη σύμβαση, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι κανόνε στην ένα οδηγία περιορίζονται από τη σύμβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, τμήμα, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρο τη ε, σύμβαση. δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα στα μισά κρατημέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια άλλα στα άλλα. Ε, με βάση το άρθρο 14. Εδώ δεν ρυθμίζονται θέμα ευθύνη. Η οδηγία για, τα, για την ασφάλεια στο άρθρο 3 λέει ότι η ευθύνη ε, ρυθμίζεται με βάση το δίκαιο του κάθε κράτου. Επομένω, το θέμα τη αποζημίωση ε, τίθεται και οι απαντήσει δεν είναι καθόλου σίγουρε. Η διάταξη λέει ότι η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει, ε, αποζημιώνει με βάση το δίκαιο του κράτους που έχει καταχωρηθεί το αυτοκίνητο ε, είτε ε, του κράτους που έγινε το ατύχημα. Στην περίπτωσή μας, αν το γερμανικό δίκαιο ισχύσει και όχι το δίκαιο του Λουξεμβούργου, οι ζημίες που δίνονται με βάση το γερμανικό δίκαιο ξεπερνούν τα όσα δίνει ο ασφαλιστής με βάση το Λουξεμβούργιο δίκαιο, ο ασφαλιστής θα πρέπει παρόλα αυτά να καλύψει το υψηλότερο κόστος με βάση το γερμανικό δίκαιο. Λαμβάνοντας υπόψη ε, την ε, ε, υψηλή προστασία που εξασφαλίζει η οδηγία για τα θύματα και που έχει επιβεβαιωθεί από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορεί ο ενάγων να καλύπτεται από την καλύτερη εκδοχή των δύο σενάριων. και θα δούμε στο παράδειγμά μας, ας πούμε, ε, το Λουξεμβούργιο δίκαιο ισχύει για την ευθύνη, ενώ το γερμανικό δίκαιο αφορά την ρυθμή στα θέματα της αποζημίωσης. Υπάρχουν πάντως αβεβαιότητες εδώ. Η αβεβαιότητα είναι σημαντική ε, και επομένως δεν ξέρουμε ποιο είναι το συμπέρασμα. Το, το τελικό συμπέρασμα είναι λίγο παράδοξο το εφαρμοστέο δίκαιο τελικά θα καθοριστεί από τη Σύμβαση της Χάγης. Αυτό ε, είναι υπέρ του, του εναγόμενου. Το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να επηρεαστεί και από την οδηγία για την ασφάλεια των αυτοκινήτων που έχει υψηλή προστασία ε, για τα θύματα. Ε, το ρόμι 2 επίσης επισέρχεται εδώ και ο κανονισμός ε, βρίσκεται κάπου ανάμεσα, στα δύο, ε, ανάμεσα στην οδηγία και στη σύμβαση και προσπαθεί να εξορροπήσει τα συμφέροντα και των δύο ε, μερών. Η περιπλοκότητα και η αβεβαιότητα είναι και μεθοδολογική και πρακτική. Απλώς άγγιξα την κορφή του παγόβονου που απορρέει από την παράλληλη ύπαρξη αυτών των εργαλείων. Γι' αυτό θα πρέπει να να τροποποιηθεί η κατάσταση. Με βάση τις πληροφορίες που έχουν δοθεί για τη δυνατότητα των θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων να ζημιωθούν από την εφαρμογή ενό ξένου δικαίου κατά την άσκηση αγωγή, ο καλύτερο τρόπο για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα είναι να βασιστούμε στην, στα μέτρα προστασία ε, των θυμάτων, στην ε, οδηγία ε, για την ασφάλεια των οχημάτων και να του δίνουμε τη δυνατότητα να μηνύουν στο χώρο συνήθω κατοικία. Έχω ετοιμάσει κάποια πληροφοριακά στοιχεία στο σημείωμα και η πρόταση αυτή που κάνω εγώ είναι παρόμοια με τον καθηγητή του κ. Στόντιγκερ. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι αν το σενάριο που σας έδωσα στην αρχή σας φάνηκε λίγο περίεργο, έχω να σας πω ότι σε λίγες εβδομάδες εγώ ακριβώς αυτό το ταξίδι θα κάνω, και αν, αν και θα ξεκινήσω από την Αγγλία, όχι από τη Γαλλία. Και με βάση ε, το τι μπορεί να με περιμένει, σας παρακαλώ να μου ευχηθείτε καλή τύχη. Σας ευχαριστούμε κυρία Παπέτας. Η ομιλία της κυρίας Παπέτας ήταν ε, η τελευταία παρουσίαση του πρωινού τμήματος ε, του εργαστηρίου μελέτης μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την έλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την παρουσίαση των πολύ ε, σημαντικών αυτών ε, και διαφορετικών παρεμβάσεων. Και μάλιστα οι εμπειρογνώμονε μα, οι καλεσμένοι μα είναι στη διάθεσή σα. Αν έχετε ερωτήσει ή σχόλια ή παρατηρήσει, ε, είναι η ευκαιρία να τα διατυπώσετε. Ποιο θέλει το λόγο. Ich möchte mich den Vorschlägen... Θα ήθελα να συμφωνήσω με τις προτάσεις αυτών των δύο εμπειρογνωμόνων τα δύο τελευταία χρόνια επανειλημμένα ως καθηγητής του Πανεπιστήμιου της, Νίρεμβέργης, της Χάιντελβέργης είδα περιπτώσεις ε, ατυχημάτων όπου συμμετέχουν άτομα από διάφορα κράτη. Κάθε φορά το θέμα είναι η, α, η απευθείας απέτηση και κάθε φορά μας ρώτησαν εμάς ποιο δίκαιο πρέπει να χρησιμοποιηθεί Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία. Η ερμηνεία σε αυτές τις περιπτώσεις, ο καθορισμός του, ποιο δίκαιο πρέπει να ε, ε, χρησιμοποιηθεί ε, κοστίζει πάρα πολλά χρειαζόμαστε καλούς εμπειρογνώμονες παίρνει πάρα πολύ χρόνο παίρνει μεταξύ 6 και 9 μηνών 6 και 9 μήνες αυτό πρέπει επίσης να πούμε ανοιχτά είναι πολύ συχνά μια διαδικασία ιδιαίτερα περίπλοκη να καθορίσουμε ποιο δίκαιο πρέπει να εφαρμοστεί Όλες αυτές είναι μη απαραίτητες διαδικασίες. Γι' αυτό υποστηρίζω πλήρως αυτή την πρόταση και ευχαρίστω. Ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι που, ε, στους οποίους τίθενται όπως και σε εμά τέτοιου τύπου ερωτήματα ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην κολονία όπου γίνονται πολλά ατυχήματα υποβάλλονται 30 με 40 τέτοια ερωτήματα κάθε χρόνο και είναι μόνο για τη Γερμανία που έχω στοιχεία, το θέμα αυτό τίθεται και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη. Όμως πρέπει να εκφράσω μία επιφύλαξη. Με αυτή την ε, χρήση ε, εφαρμογή ε, του δικαίου της χώρας όπου διαμένει συνήθως το άτομο δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Συνάδελφοι από την κολονία, που πολλές φορές έχω κληθεί ως εμπειρογνώμονες να διευκρινίσουν αυτά τα δύσκολα ερωτήματα, για παράδειγμα ε, ποιο είναι το όριο ταχύτητα για φορτηγά ε, στην Ολλανδία. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα, αλλά παρόλα αυτά καλωσορίζω την πρόταση. Σας ευχαριστούμε καθηγητά Χες για τι παρατηρήσεις. Όσο περισσότερα κενά υπάρχουν, τόσο περισσότερα παραθυράκια ανοίγουν για τέτοιου είδου φαινόμενα που είναι κυρίως επιβλαβή και επιζήμια για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό δεν θέλουμε να θεσπίσουμε δίκαιο που θα διευκολύνει ε, τη ζωή όλων μας και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο επίπεδο. Θέλει άλλος κανείς το λόγο, παρακαλώ. Ε, ε Μήπως θα μπορούσε πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να λάβει το λόγο. Κυρία Μίχου. I fully Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και φέτος και του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει ενδελεχώς όλα αυτά τα θέματα που ακούσαμε προηγουμένως και φυσικά δεν μπορώ να προδικάσω την έκβαση αυτής της ε, εξονυχιστικής μελέτης, αλλά πιστεύω ότι στη διάρκεια της συζήτησης αυτής και της εξέτασης αυτής θα δημιουργήσουμε τη βάση και τα θεμέλια για τις μελλοντικέ μας αποφάσεις. Ε, αυτό είναι το πρόγραμμα και ο σκοπός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχαριστώ όλους όσους λάβατε μέρος σε αυτό το πρωινό τμήμα του σεμιναρίου μας και αν δεν θέλει άλλο το λόγο μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας του πρώτου μέρους και να δώσουμε ραντεβού και πάλι για τις 3 με την αναρκτήρια ομιλία του πρώην συναδέλφου Κουρτ Λέχνερ που είναι γνωστός και αγαπητός σε όλους. Το δεύτερο μέρος λοιπόν θα αρχίσει στις 3 ε, και στις 5 το τρίτο μέρος του σεμιναρίου. Σας ευχαριστώ και τα ξαναλέμε το απόγευμα στις 3. work.